Buenas Καλησπέρα. Estar presidida esta comisión δε hoy. Σήμερα θα προεδρεύσω εγώ στα Ισπανικά. Ζητώ καταρχά συγγνώμη η κυρία Χολμάγερ, διότι δεν θα μπορέσει να βρεθεί σήμερα εδώ μαζί μα. Θα περάσουμε λοιπόν απευθεία στην ημερήσια διάταξη. Έχετε λάβει το σχέδιο ημερήσια διάταξη στι 25 Οκτωβρίου του 2019. Επομένως, αν δεν υπάρχουν ενστάσει, εγκρίνετε. Υπάρχει κάποια αντίρρηση, συμφωνείτε. Ωραία, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Όπως γνωρίζετε όλες εσείς, υπάρχει διερμηνία σε 14 γλώσσες. Να καλωσορίσουμε τους διερμηνείς και να τους ευχαριστήσουμε που μας επιτρέπουν να μπορούμε να εκφραστούμε στην μητρική μας γλώσσα και να το υπενθυμίσω και στους ευρωβουλευτές ότι υπάρχει διαθέσιμη όλη η τεκμηρίωση της συνεδρίασης και της σημερινής ε, συνάντησης στην ε, ιστοσελίδα ε, της ΚΟΝΤ. Έγκριση των συστάσεων των συντονιστών τη συνεδρίαση που έγινε στις 8 Οκτωβρίου του 2019 με τις συστάσεις. Έχουμε μία σύνοψη ε, και επομένως ε, εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις μέχρι το πέρας της συνεδρίασης θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται και τα πρακτικά και οι συστάσεις των συντονιστών. Περνάμε τώρα στην έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων για τις ε, 25 και 26 Σεπτεμβρίου και 8 και 17 Οκτωβρίου. Τα στείλαμε όλα στις 7 Νοεμβρίου. Αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, εγκρίνονται τα πρακτικά. Έχει κάποιος κάτι να πει. Εγκρίνονται λοιπόν και τα πρακτικά. Και περνάμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης για τις διαπραγματεύσεις για ε, την Όλαφ. Ο κύριος Μαρινέσκου είναι ο εισηγητής. Ο πρώτος διοργανικός ε, τριμερής διόλογος έγινε στις 7 ε, Νοεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βάσει του άρθρου 74 προβλέπεται στην επόμενη συνεδρίαση να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ενημερωθεί η Επιτροπή μας Δεν είναι εδώ. Ο κύριος Μαρινέσκου λοιπόν απουσιάζει. Δεν ξέρω αν έρθει αργότερα, θα μπορούσαμε ίσως να του δώσουμε το λόγο. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 5 στη συνέχεια. Απαλλαγή 2018, Γενικός Προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο τον κύριο Αβραμόπουλο Επίτροπο Αρμόδιο για τη Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια, τον οποίο καλωσορίζω θερμά και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την διαθεσιμότητά του να συναντηθεί με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τον κύριο Μπρίνκα, το οποίο είναι μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στείλαμε ένα κατάλογο ερωτήσεων στον Επίτροπο οι απαντήσεις έχουν δοθεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Ε, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, λοιπόν, να δώσω το λόγο στον κύριο Μπρίνκατ για να μας παρουσιάσει ε, τις εντυπώσεις του εντός 10 λεπτών. Κύριε Μπρίνκατ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε. Κυρίες ε, και κύριοι βουλευτές ε, και κύριοι επίτροπες, σήμερα εκπροσωπώ εδώ το ελεγκτικό συνέδριο όσον αφορά το κεφάλαιο 8 της ετήσιας έκθεσης του για το οικονομικό έτος 2018. Για τρίτη συνεχή χρονιά έχουμε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για την ασφάλεια και την ηθαγένεια στην ετήσια έκθεσή μας, το οποίο αφορά την ομότητα και κανονικότητα των δαπανών της Ένωσης. Τα ευρήματα σε αυτόν τον ε, τομέα εντάσσονται στα γενικότερα συμπεράσματά μας για τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν κάνουμε όμως μια συγκεκριμένη αξιολόγηση για τον τομέα αυτών των δαπανών, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 2% του συνολικού κοινοτικού προπολογισμού. Για το 2018 οι δαπάνες ήταν γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ στον τομέα αυτών. Παρ' όλα αυτά, το ελεκτικό συνεδρίο αναγνωρίζει το ενδιαφέρον των πολιτικών και του κοινού σε αυτόν τον τομέα που είναι πολύ υψηλότερο από το ποσοστό της χρηματοδότησης. Γι' αυτό αποφασίσαμε να μην ελέγξουμε μόνο τις ε, συναλλαγές, αλλά να δούμε και τα συστήματα ελέγχου και τη λειτουργία της διοίκησης των κρατών μελών και της Γενικής Διεύθυνσης ε, της ε, Κομισιόν επιπλέον εξετάσαμε την απόδοση κάποιων βασικών πτυχών των πολιτικών μετανάστευσης της Ένωσης. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε στις εκθέσεις μας όπως η SR 20-2019 για τα πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζουν τον έλεγχο των συνόρων, η SR 24-2019 για άσυλο με την κατάσταση και επιστροφές που θα δημοσιευτεί την Πέμπτη και για την οποία επίσης αντιλαμβάνομαι ότι έχει προγραμματιστεί τον επόμενο μήνα μια συνεδρίαση με την Επιτροπή σας και επίσης η ε, δουλειά που κάνουμε για την Frontex, ε, για την οποία είμαι επίσης εισηγητής. Η δουλειά μας ε, για το 2018, η έκθεσή μας, αποκάλυψε ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο καλύτερης χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων σε αυτό το ΠΔΠ διασφαλίζοντας παραδείγματο χάρη ότι τα κράτη-μέλη θα ε, εκταμιεύουν μόνο όταν πληρούνται όλοι οι όροι, όταν γίνεται έλεγχος μετά από έλεγχο όλων των κριτηρίων επιλογής χαιρόμαστε για το ότι ο βαθμός εφαρμογής των προγραμμάτων έχει αυξηθεί σημαντικά και η Κομισιόν έκανε περισσότερες δαπάνες το 2018 από όσο συνολικά τα προηγούμενα τρία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, στο υφιστάμενο πλαίσιο μεταναστευτικών πιέσεων και απειλών ασφαλείας, τα κράτη-μέλη δεν εξαντλούν τα κοινοτικά κονδύλια που υπάρχουν στην διάθεσή τους για να διαχειριστούν τις μεταναστευτικές ροές και να ενισχύσουν τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων μας. Κατανοητό είναι ότι τα κονδύλια τα οποία δεν έχουν ξοδευτεί, συνεχίζουν να αυξάνονται και θα αυξηθεί επίσης τα εθνικά συστήματα προς το τέλος του ΠΔΠ. Το κεφάλαιο 2 της έκθεσής μας επίσης αναφέρεται στον αντίκτυπο που έχουν οι καθυστερήσεις αυτές. Ο έλεγχος των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδια για την εφαρμογή των προγραμμάτων MFISF δείχνει πως ε, έχουν ε, ενισχύει επαρκείς ελέγχους για την εφαρμογή αυτών των κανονισμών. Το ίδιο ισχύει και για τις εσωτερικές διαδικασίες της Γενικής Διεύθυνσης ε, Home για την αξιολόγηση των επιχορηγήσεων και την εξοδότηση των πληρωμών. Όταν είδαμε ότι χρειαζόταν κάποιες βελτιώσεις, σε σχέση δηλαδή με την επαλήθευση των δαπανών ή τον έλεγχο των διαδικασιών δημοσίων προμηθειών και επιλογής, κάναμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις οι οποίες σε γενικέ γραμμές έγιναν δεκτές από τις εθνικές αρχέ. Όσον αφορά την απόδοση, η δουλειά που γίνεται στα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιεί πάντα τους απαραίτητους δείκτες στο κατάλληλο επίπεδο στο αποτέλεσμα αυτού. Λυπούμαστε για το ότι ο αντίκτυπο των έργων αυτών δεν μπορεί να μετρηθεί επακριβώς υπό αυτές τις συνθήκες. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και τη Γενική Διεύθυνση Home για το επίπεδο της συνεργασίας που έχουν επιδείξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο. Παρακαλώ, κύριε Βραμόπουλο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που βρίσκομαι και πάλι εδώ και να ευχαριστήσω και πάλι και εσάς και όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Χαίρομαι που βρίσκομαι και πάλι στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Δεν είναι η πρώτη φορά και το ξέρετε πολύ καλά. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και τον κύριο Μπρινκάτ για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. και είμαι βέβαιος ότι στη σημερινή συνεδρίαση θα μπορέσουμε να ρίξουμε λίγο φως σε όλες τις πτυχές οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη διαχείριση των πιο σημαντικών θεμάτων των τελευταίων πέντε ετών. Σήμερα έχουμε ανοιχτή συζήτηση για τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2018 και στον τομέα της μετανάστευσης και στον τομέα της ασφάλειας. Όπως γνωρίζετε, αυτή είναι η τελευταία φορά που θα ε, μιλήσω εδώ στην Επιτροπή σας και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία να συνοψίσω την πρόοδο που επιτύχαμε την τελευταία πενταετία και πιο συγκεκριμένα το 2018. Στη διάρκεια της τελευταίας ε, πενταετίας, πιστέψτε με, προσπαθήσαμε να βρούμε τις καλύτερες δυνατές και τις πιο βιώσιμες λύσεις, προκειμένου να βοηθήσουμε όσους χρειάζονται διεθνή προστασία, να μειώσουν να μειώσουμε τα κίνητρα για την ε, παράτυπη μετανάστευση και να διαχειριστούμε καλύτερα και να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας ε, σύνορα, καθώς επίσης και να δημιουργήσουμε ασφαλείς και νόμιμες ε, οδούς. Ακριβώς λοιπόν υπό αυτό το πνεύμα θέσαμε και τα θεμέλια για μια συνολική ε, πολιτική μετανάστευση η οποία ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις ε, και βασίζεται αποτελέσματα στην αλληλεγγύη και στην ευθύνη. Ταυτόχρονα προτείναμε και μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ασφάλεια για να έχουμε μια αποτελεσματική ένωση ασφαλείας. Βεβαίως ε, μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι ακόμα μας περιμένει πολλής δρόμος, αλλά το 2018 συνεχίσαμε να παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για την επίτευξη αυτών των στόχων. Να ξεκινήσω τώρα με τη μετανάστευση. Το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πολύ συγκεκριμένε προτάσεις ε, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση για να προστατεύσει καλύτερα τα εξωτερικά της σύνορα δίνοντας ε, μια αυξημένη νομοθεσία για την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Λιμενοφυλακή και ένα μόνιμο προσωπικό περίπου 10.000 συνοριοφυλάκων. Αυτό θα υλοποιηθεί από το Δεκέμβριο φέτος με την έναρξη ισχύω ε, του νέου κανονισμού. Και φυσικά ενίσχυση των ε, επιστροφών μέσω μιας αναδιατύπωσης της οδηγίας για τις επιστροφές. Ταυτόχρονα θέλουμε να ενισχύσουμε τις νόμιμες οδούς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξυγχρονίσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες θεωρήσεων διαβατηρίων με πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας του κώδικα των θεωρήσεων, κάτι το οποίο έχουμε ήδη ε, εγκρίνει και σε επίπεδο VIS, του συστήματος, ε, ε, πληροφορικού συστήματος των θεωρήσεων. Αυτό θα βοηθήσει για αποτελεσματική διαχείριση των σύνορων. Η γρήγορη εφαρμογή φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντική για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Τα στοιχεία του 2018 αντικατοπτρίζουν τα απτά αποτελέσματα των συνεχών προσπαθειών μας και πιο συγκεκριμένα τον αριθμό των παράτυπων διελεύσεων των συνόρων που μειώθηκαν και έφτασαν σε επίπεδα πριν από την κρίση. Πάνω από 25.000 από τους πιο ευάλωτες ε, μετανάστες επανεγκαταστάθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την υποστήριξη ε, κονδυλίων από την ε, Γενική Διεύθυνση Home, έτσι, με τα κονδύλια αυτών είχαμε σημαντική ε, χρηματοοικονομική υποστήριξη προς τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων. Από το 2016 και μέχρι τώρα η Ελλάδα έχει λάβει 2,2 δις ευρώ για την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης και των συνόρων, ενώ η Ιταλία εποφελήθηκε από περίπου ένα δις ευρώ. Και η στήριξή μας συνεχίζεται. Επιπλέον, το 2018 το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης υποστήριξε τα κράτη-μέλη για την επιστροφή περίπου 40.000 ατόμων σε σύγκριση με τα 16.000 άτομα που είχαμε το 2017. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, έχουμε ακόμα πάρα πολλή δουλειά. Πιο συγκεκριμένα, ενώ έχουμε επιτύχει σημαντική πρόοδο, δυστυχώς τα κράτη-μέλη δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα σύλλου όπως είχαμε προτείνει. Χρειαζόμαστε κατεπηγόντως ε, μία εις βάθος ε, μεταρρύθμιση των κανόνων ε, ασύλου καθώς επίσης και ισχυρότερα εξωτερικά σύνορα, γεγονός το οποίο θα μας επιτρέψει να διαχειριστούμε οποιαδήποτε μελλοντική πρόκληση συλλογικά και με δίκαιο τρόπο. Υπ' αυτό το πλαίσιο βασίζομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υποστηρίξουμε τις μελλοντικέ εργασίες για ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, όπως ε, ανακοινώθηκε και από την ε, ε, εκλεγμένη πρόεδρο. Το περιεχόμενο της πολιτικής μας ε, ήταν ανέκαθαν η στρατηγική εταιρική σχέση με τρίτες χώρες και ένα από τα βασικά παραδείγματα είναι η συνεργασία με την Τουρκία βάσει των δηλώσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ε, που το 2018 συνέχισαν τη μείωση των παράτυπων μεταναστών και μειώθηκε και ο αριθμό των ε, ζώων που χάνουμε στη θάλασσα. Επαναλαμβάνω στους τουρκούς εταίρους ε, και το επανέλαβα και στην πρόσφατη επίσκεψή μου στην Άγκυρα τον περασμένο μήνα ότι πρέπει να συνεχίσει η δέσμευση και η συνεργασία μας. Επιτρέψτε μου τώρα να περάσω σε, στην ασφάλεια. Οι επονίδε στι τρομοκρατικέ επιθέσει που αντιμετώπισε η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια κατέδειξαν ότι χρειαζόμαστε ένα συνολικό, ευρωπαϊκό και διεθνέ ε, ε, σύστημα για την αντιμετώπιση των απειλών ασφαλεία. Το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μία σειρά από νομοθετικέ προτάσει για την αντιμετώπιση τη τρομοκρατία και του οργανωμένου εγκλήματο με στόχο την ενίσχυση των κανόνων για την εμπορία και τη χρήση ε, εκρηκτικών και πρόδρομων ουσιών, ε, τη διευκόλυνση των πληροφοριών που αφορά ποινικά αδικήματα και ε, τα κατάλληλα εργαλεία προς τις εθνικές αρχές για την αντιμετώπιση και έρευνα εγκληματικών πράξεων με σύγχρονα μέσα. Το έργο μας δεν σταμάτησε εδώ. Η αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Και ενώ καταφέραμε να κερδίσουμε το ISIS ε, επιτόπου, το διαδίκτυο έχει γίνει ε, το πιο σημαντικό πεδίο μάχης. Αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέψαμε το 2015, όταν ανέλαβα την πρωτοβουλία για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Διαδικτυακού Φόρουμ. Το 2018 κάναμε ένα βήμα παραπέρα και προτείναμε Πανευρωπαϊκού κανόνες ε, για την πρόληψη της δημοσιοποίησης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Χαίρομαι που ξεκίνησε πρόσφατα ο τριμερής διάλογος ε, και είμαι βέβαιος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμβάλλει στην ε, γρήγορη έγκριση αυτής της πρότασης. Επίσης, εργαζόμαστε για να ε, μειώσουμε τα κενά στις πληροφορίες ε, και να μπορέσει να υπάρχει και συνεργασία των πληροφοριακών συστημάτων. Τα κράτη-μέλη από την πλευρά τους πλέον πρέπει να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των νέων κανόνων. Όλες αυτές οι δραστηριότητες για τη μετανάστευση και την ασφάλεια διέπονται από αυξημένο προπολογισμό στο πρόγραμμα ε, του πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου. Γεγονό το οποίο μα επιτρέπει να υποστηρίξουμε τι προσπάθειε και τι προτεραιότητέ μα ε, με συγκεκριμένη ε, ασφάλεια και με πολύ στοχευμένο αριθμό ε, επιφυλάξεων. Όσον αφορά τα απορίσματα του ελεκτικού συνεδρίου, με χαρά διαπιστώνω ότι το ελεκτικό συνέδριο δεν έχει διαπιστώσει να υπάρχει μεγάλη ε, διαφορά και προβλήματα στην εφαρμογή, ούτε στο Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, ούτε στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας. Όπως παρατήρησε το δικαστήριο το 2018, τα κράτη-μέλη έχουν αναβαθμίσει την εφαρμογή των εθνικών τους προγραμμάτων και τώρα περιμένουμε αυτή η θετική ε, τάση να συνεχιστεί. Επίσης είμαι ικανοποιημένος από τη δήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου ότι οι εσωτερικές διαδικασίες της Γενικής Διεύθυνσης Home για, τις, ε, για την έγκριση των αιτήσεων ενίσχυσης και των εσωτερικών διαδικασιών είναι ε, σωστές και σωστά τεκμηριωμένες. Οι μηχανισμοί εσωτερικών ελέγχων και ε, επιθεωρήσεων λειτουργήσαν επίσης καταλήλω και αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι μόνες αδυναμίες που εντόπισε το, δικαστήριο σε σχέση, το ελεγκτικό συνέδριο σε σχέση με την Ισπανία είχαν ήδη αντιμετωπιστεί πριν γίνει εκαθάριση ή έγκριση για οποιαδήποτε λογαριασμό. Η ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ε, διαπιστώνει ότι υπήρξε καλή πρόοδος για αποτελεσματική εφαρμογή των ε, ταμείων και σεβόμενη επίσης και τα θέματα της χρηστής οικονομικής διαχείρισης. Χαίρομαι για την ε, ε γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις υπόλοιπες πέντε υπηρεσίες και οργανισμού μας για το 2018. Θα αναφερθώ τώρα ε, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Στήριξης ε, ε, του Ασύλου. Όλοι γνωρίζουμε πως το ΕΑΖΟ έχει αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις στο παρελθόν και θα χρειαστεί χρόνος μέχρι ότου ενισχυθεί πλήρως το πλαίσιο εσωτερικής διακυβέρνησης να αποκατασταθεί η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη. Ωστόσο όλοι συμφωνούμε ότι τα μέτρα που χρειάζονται για να βελτιωθεί, μάλλον που για να βελτιωθεί η διακυβέρνηση του του οργανισμού αυτού έχουν ήδη επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Η επόμενη ε, ε, διευθύντρια που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούνιο του 2019 ε, η κυρία Νίνα Γρηγόρη θα εξασφαλίσει την εφαρμογή όλων των συστάσεων ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αξιοπιστία της ΕΑΖΟ. Είμαστε, εξακολουθούμε να στηρίζουμε το πρόγραμμα δράσης ε, που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2018, διότι δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί αυτό το έργο, όπως φαίνεται και από την γνωμοδότηση του ε, δικαστηρίου. Εμείς ε, παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ στενά ώστε να εξασφαλίζουμε ότι ο οργανισμός θα ακολουθεί τις συστάσεις του ελεγκτικού συνέδριου όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά και όσο γίνεται και πιο γρήγορα. Τώρα, αν δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις στον τομέα του ασύλου, η Κομισιόν υπέβαλε πρόταση το 2016 για μετατροπή της ΕΑΖΟ σε πλήρη οργανισμό, ευρωπαϊκό οργανισμό ασύλου, ώστε να, έχει καλύτερα, να είναι καλύτερα εξοπλισμένος ο οργανισμός αυτός για να πληρεί αυτό την εντολή. Επίσης, το 2016 η Κομισιόν πρότεινε να ενισχυθεί περαιτέρω η ΆΖΟ, ώστε να εξασφαλίσουμε πως θα παρέχει στα κράτη-μέλη όλη την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη. Σας καλώ εσάς και τα κράτη-μέλη, ώστε να εξασφαλίσουμε την ε, ταχεία έγκριση αυτής της πρότασης. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, η χρηματοδότηση για την μετανάστευση και το άσυλο έχει εξυπηρετήσει τις πολιτικές που ωφελούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι πολίτες ε, και δικαίως αναμένουν λύσεις από πλευράς μας και αυτό είναι σημαντικό να εφαρμόσουμε αυτές τις πολιτικές και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Επί τόπου. Για να το καταφέρουμε αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε κατάλληλη χρηματοδότηση αυτών των πολιτικών και στα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό το στόχο βασίζομαι και στη στήριξη ε, του δικού σας σώματος ε, που έχει εκφραστεί ε, στο παρελθόν επανελειμμένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη σας την υποστήριξη, για την υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων στον τομέα της ασφάλειας που αντιμετωπίζει τόσο μεγάλες προκλήσεις. Ε, οι αξίες μας που μας ενώνουν, μας ενώνουν όλους και διέπουν τις εργασίες μας τον τελευταίο, την τελευταία πενταετία. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτή το κληροδότημα. Ελπίζω πως αυτή η εξαιρετική συνεργασία και εμπιστοσύνη θα συνεχιστεί και στο μέλλον και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής, ξεκινώντας ε, από την κυρία Winfield που αντικαθιστά την κυρία Χόλμαϊερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν εξ ονόματος της ε, κυρίας Χολμάιερ το το μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά και την ε, Κομισιόν για τις απαντήσεις της. Ε, η κυρία Ολμαϊρ όμως έχει κάποιες ερωτήσεις. Δεν βλέπουμε εδώ πέρα πότε ανατέθηκαν οι μελέτες και πότε δημοσιεύτηκαν. Επιπλέον ε, δεν ξέρουμε αν χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των μελετών αυτών και ποια συγκεκριμένα μέτρα ελήφθησαν. Επίσης δεν δημοσιεύτηκαν οι πέντε μελέτες που αναφέρονται. Στην απάντηση της ερώτησης 16 η Κομισιόν λέει ότι οι ελληνικές αρχές ε, προσπαθούν ε, να βγάλουν τα συνοδευτά ανήλικα το συντομότερο δυνατόν από το hotspot. Ε, υπάρχουν όμως μεγάλα προβλήματα εδώ πέρα η Κομισιόν περιγράφει θετικές εξελίξεις στα Ιταλικά hot spot όπου η μέση διάρκεια παραμονής των ανηλίκων έχει μειωθεί σημαντικά. Μπορεί η Κομισιόν ε, να μας πει αν έγιναν βελτιώσεις και στην Ελλάδα και πώς έχει η κατάσταση σε Ελλάδα και Ιταλία σε σχέση με άλλους ε, ευπαθείς ε, όπως παραδείγματος χάρη ανάπηρους ή εγγύους για τις επιστροφές ε, τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν για το ότι στην Ελλάδα άτομα που δεν δικαιούνται άσυλο δεν ε, απελάβνονται από την χώρα σύμφωνα με την συμφωνία με την Τουρκία. Ποια μέτρα θα λάβει η Κομισιόν έτσι ώστε να μην υπάρχει κατάχρηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων με αυτόν τον τρόπο και να βοηθούνται πραγματικά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη. Ποια είναι η αιτία των προβλημάτων αυτών για την ε, κατάχρηση, όπως είπα, των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων για λάθος σκοπούς. Τέλος, για την τεχνική αρρωγή. Θεωρεί η Κομισιόν ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω τεχνική αρρωγή για τις τοπικές αρχές. Και στην απάντησή σας στο ερώτημα 24 λέτε ότι υπάρχει μία ανάγκη ανάκτησης ε, αχρεωστήτων καταβληθέντων αμφισβητήθηκε αυτό από κάποιο κράτος μέλος και πώς ακριβώς θα τα ζητήσει αυτά τα λεφτά η Κομισιόν πίσω και πότε υπολογίζει να ανακτήσει ολόκληρο το ποσό. Κατά ποιον κρατών μελών απευθύνονται αυτές οι εντολές ανάκτησης ε, χρημάτων. Θα πρέπει η Κομισιόν να μας πει σε ποια κράτη-μέλη και για ποια ποσά και για ποιον λόγο. Μετά η κυρία Χολμάιρ έχει κάποιες ερωτήσεις ε, προς το ελεγκτικό συνέδριο για την τεχνική αρρωγή. Θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη για βελτιώσεις ε, και επέκταση της ε, τεχνικής αρρωγής. Θα μπορούσε στο πλαίσιο αυτό το ελεγκτικό συνέδριο να μας πει αν υπήρξαν βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια και πού βλέπετε ότι υπάρχει περιθώριο για απλοποίηση των κανονισμών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στους ε, σκιώδεις εισηγητές. Ξεκινούμε με την κυρία Πίνκοβα από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε και ευχαριστώ κυρία Βραμόπουλε. Φυσικά τα όσα μας λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικά και γι' αυτό και οι πληροφορίες που μας δίνετε σήμερα είναι ε, κέριο ενδιαφέροντος για όλους μας εδώ. Έχω δύο ερωτήσεις ε, για σας. Η πρώτη σχετίζεται με την μικρή απορρόφηση του κονδυλίου μετανάστευσης και του κονδυλίου για την εσωτερική ασφάλεια που αναφέρατε. Τι κάνει η Κομισιόν για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν το ποσοστό απορρόφησης για αυτά τα κονδύλια. Συγκεκριμένα δηλαδή τι βοήθεια προσφέρεται στα κράτη-μέλη. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά την εργασία των έξι αποκεντρωμένων οργανισμών που στηρίζουν την εργασία της DigiHome. Θέλω δηλαδή να καταλάβω πώς συντονίζει η Κομισιόν την εργασία αυτών των οργανισμών, πώς αποκομίζεται διδάγματα από την εκτέλεση των προπολογισμού και των πολιτικών που θα μπορέσετε να μοιραστείτε με άλλους οργανισμούς και θα αποφύγετε ε, σφάλματα την επόμενη χρήση. Ευχαριστώ πολύ. Señor Chastel, por Ευχαριστώ από το Ρινιού Σαστέλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Καταρχά να σα ευχαριστήσω πολύ για την παρουσίαση τη έκθεση δραστηριοτήτων τη DG Home, πράγμα που συμπληρώνει τα όσα λάβαμε από το ελεγκτικό συνέδριο και την έκθεση για το 2018 για τη διαχείριση και την απόδοση του προπολογισμού τη Ένωση. Είναι αλήθεια ότι η DG μετανάστευση αντιπροσωπεύει μόνο το 2% του προπολογισμού. Είναι όμω μία από τι πιο συμβολικές ε, διευθύνσει σε σχέση με τις πολιτικέ που ασκούνται, ιδιαίτερα με την κρίση των Συρίων μεταναστών, την κατάσταση της Μεσογείου, τη σημασία ασφάλισης των εξωτερικών συνόρων, την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευση, την δημιουργία μια αξιόπιστη πολιτικής και μια εναρμονισμένης πολιτική για θέματα ασύλου και μετανάστευση. Αυτέ τι αποστολέ φυσικά θα πρέπει να τις συνεχίσουμε και σε αυτή τη θητεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να δώσει λύσεις και από αυτό εξαρτάται η αξιοπιστία της. Η ετήσια έκθεση της Κομισιόν ε, προτάσει ότι η ΔΕΖΕ έχει γενικά διαχειριστεί καλά το κονδυλιά τη και τα αιτήματα επιδοτήσεων και όλα αυτά, όμως μένουν κάποια κενά στην εφαρμογή των κανόνων της, των δημόσιων ε, ε, κρατικών διαγωνισμών αλλά και στη διαχείριση των χρημάτων για το άσυλο και τη μετανάστευση και για την εσωτερική ασφάλεια που είναι κοινή διαχείριση με τα κράτη. Κύριε Επίτροπε, στην έκθεση δραστηριοτήτων η Γενική Διαθήση λέει ότι το ποσοστό απόδοσης είναι εν γέννη 41,8% και 35,63% προς τις τρίτες χώρες πιο συγκεκριμένα. Αυτά τα νούμερα είναι προς τα κάτω, είναι καθοδικά το 2016, από το 2016 και σημαντικά κονδύλια αφιερώνονται. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή προβλέπονται για να αυξηθούν αυτά τα νούμερα που είναι πολύ χαμηλά εδώ και χρόνια παρά τους προϋπολογισμούς που δίνονται. Πού βρίσκονται οι συμφωνίες επανεισδοχής με τις χώρες του Μαγκρέμπου που η Κομισιόν έχει λάβει την εντολή των κρατών μελών εδώ και χρόνια. Επίσης τι συμβαίνει με τις χώρες του Σαχέλ. Άλλη ερώτηση. Το ελεγκτικό συνέδριο διαπιστώνει πως ε, ε, τα κονδύλια που δεν έχουν δαπανηθεί αυξάνονται, πράγμα που σημαίνει αύξηση των επιστροφών προς τα κράτη εφόσον ολοκληρώνονται τα μέτρα. Ε, τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Έπειτα, στην δήλωση ε, ασφάλισης. Ε, το δικαστήριο δείχνει κάποια προβλήματα όσον αφορά την υιοθέτηση των προγραμμάτων και την αξιολόγηση των επιδοτήσεων και ζητά καλύτερο έλεγχο στις διαδικασίες. Ποια μέτρα λοιπόν έχουν ληφθεί συγκεκριμένα ώστε να αυξηθεί η απόδοση των προγραμμάτων και η νομιμότητα και η κανονικότητα των ε, δημοσίων διαγωνισμών. Ποια είναι τα μέτρα που ελήφθησαν να αυξηθεί η χρήση των δικτών απόδοσης. Επίσης θέλω να αναφέρω ε, τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν κάποια μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης ε, των χορηγιών ώστε να μειωθεί το ποσοστό σφάλματος που υπάρχει ε, σε αυτό το θέμα, των υποτροφιών με συγχωρείτε. Το σχέδιο δράσης για, κατά της, δρα, της διακίνησης μεταναστών που φτιάχτηκε το 2018 έχει εφαρμοστεί πλήρως, μπορούμε ήδη να καταμετρήσουμε θετικά στοιχεία. Τέλος, ποιον απολογισμό κάνετε εσείς από την εφαρμογή του Eurosur που διαχειρίζεται την εποπτεία των συνόρων και γενικότερα του προγράμματος Smart Borders. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πέξκα για τους πρασίνους. θα θέσετε τι ερωτήσει μου στα γερμανικά. Ε, Κύριε Επίτροπε, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να κάνω την ερώτησή μου. Το θέμα αφορά την κατάσταση στην Λιβύη. Τι κάνει η Κομισιόν για να διασφαλίσει ότι οι αρχές που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι είδου έλεγχο υπάρχει για να παρακολουθούμε την δουλειά των λιβικών αρχών και τις ε, δαπάνες επίσης ε, τις σχετικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ε, Έχουμε εκπροσώπους ε, από τις άλλες πολιτικές ομάδες και συγητές. Να δώσουμε λοιπόν και πάλι το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει στις ερωτήσεις και στα σχόλια. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχάς... Θα ήθελα να πω ότι όλες οι ερωτήσεις είναι πολύ σημαντικές. Να ξεκινήσω από τα παιδιά. Έχω επανειλημμένα πει ότι η ασφάλεια των ανηλίκων, ειδικά των ασυνόδευτων, θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα για όλους μας. Αυτό το έχουμε επαναλάβει με όλα τα κράτη-μέλη και στις ε, σχετικές αρχές και ασκούμε πίεση. Χρειαζόμαστε γρήγορη δράση. Στην Ελλάδα με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, οι αρχές έχουν αναλάβει δράση για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των ασυνοδευτών ανηλίκων στα hot spot. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης χρηματοδοτεί μέτρα για να βελτιώσει τις ε, συνθήκες διαβίωσης ε, και να βοηθήσει τους ευπαθείς ετούντες στα spot. Αλλά ναι, η κατάσταση παραμένει δύσκολη το 2019 με την στήριξή μας η Ελλάδα ανέπτυξε μια στρατηγική για τους ασυνόδευτούς ανηλίκους η οποία τώρα αναπροσαρμόζεται και κάτι το οποίο η Κομισιόν παρακολουθεί στενά σας διαβεβαίω. Επίσης αντιλαμβάνομαι ότι το Υπουργείο Προστασίας ε, του Πολίτη έχει δεσμευτεί για την γρήγορη μετακατάσταση 5.000 ανηλίκων στην Ελλάδα. Στην ε, Ιταλία οι ασυνόδευτοι ανηλικοί πηγαίνουν σε ειδικέ εγκαταστάσεις σχεδόν τη αφήξη τους τα τελευταία πέντε χρόνια. 539 δραστηριότητες που στοχεύουν ε, τα παιδιά εφαρμόστηκαν σύμφωνα με το Ταμείο Ασύλου και Ένταξης. Η συνολική κοινοτική συνεισφορά ανέρχεται σε 550 εκατομμύρια ευρώ. 50 εκατομμύρια πηγαίνουν για τις 2.000 θέσεις ε, σε ειδικέ εγκαταστάσεις για συνοδευτούς ανηλικούς στην Ελλάδα. Επιπλέον 19.000 ανηλικοί επανεγκαταστάθηκαν και 21.400 επανεγκαταστάθηκαν μεταξύ 2014 και 2018. Επιπλέον, από το 2017, η Κομισιόν και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για να στηρίξουν τα κράτη-μέλη. Έχουν επίσης οριστεί ομάδες στήριξης παιδιών σε όλα τα hot spots στην Ελλάδα. Έχει υπάρξει ένα δίκτυο αναδόχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να στηρίζει τέτοια συστήματα προστασίας παιδιών σε χώρες προέλευσης και διέλευση. Τώρα όσον αφορά τα hot spot. Η Κομισιόν συνεργάζεται στενά με τι ελληνικέ αρχές σε οικονομικό, πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο για να αντιμετωπίσει την δύσκολη κατάσταση που υπάρχει. Μάλιστα, είμαστε σε καθημερινή επαφή με μόνιμη παρουσία στην Αθήνα και στα νησιά. Ο ρόλος των εθνικών αρχών στην αντιμετώπιση της ε, κατάστασης ε, παραμένει ε, κορυφαίας σημασίας. Και βεβαίω οι ελληνικές αρχές είναι υπεύθυνες σε τελική ανάλυση. Η Κομισιόν δεν μπορεί παρά μόνο να στηρίξει και όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις ελλαδικές αρχές. Η τεράστια πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή πρόκληση. Άρα ήταν προτεραιότητα για την Κομισιόν από την πρώτη μέρα να βοηθήσει την Ελλάδα να την αντιμετωπίσει. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσουμε να παρέχουμε στήριξη στις εθνικές αρχές. Σήμερα είναι σαφές ότι απαιτείται δράση κατεπίουσα και αποφασιστική για να ανακουφιστεί η πίεση στα νησιά και να βελτιωθούν οι συνθήκες για μετανάστες και πρόσφυγες. Ο έχει στηρίξει την Ελλάδα, όπως είπα στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις, με 2,2 δισεκατομμύρια από το 2015. Τη μεγαλύτερη οικονομική στήριξη που δόθηκε ποτέ σε κράτος μέλος για τη μετανάστευση. Και τεχνικά και επιχειρησιακά. Όλοι γνωρίζουμε το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στα νησιά και δύσκολες συνθήκες ε, για τους μετανάστες. Όπως ξέρουμε, από το τέλος του Οκτωβρίου 2018 υπήρχαν ε, πάνω από 13.000 ε, παρόντες στα hot spots στα νησιά. Ο νέος ελληνικός νόμος περί ασύλου εγκρίθηκε στις 31 Οκτωβρίου. Λοιπόν, αναμένουμε την επίσημη κοινοποίηση της νομοθεσίας από τις ελληνικές αρχές Εν τω μεταξύ όμως η Κομισιόν ε, ξεκίνησε να τον εξετάζει για να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται πλήρως με το κεκτημένο. Ο στόχος παραμένει να γίνουν οι διαδικασίες πιο αποτελεσματικές χωρίς να υπάρχει ε, κάποιος συμβιβασμός για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό είναι σημαντικό για να αποσυμφορηθούν τα νησιά επιστρέφοντας αυτούς που πρέπει να επιστραφούν σύμφωνα με την δήλωση με την Τουρκία ή να μεταφερθούν ή ευάλωτοι ενήλικοι. Επίσης ε, είμαστε σε άμεση επαφή με ελληνικές και τουρκικές αρχές ε, σε πολιτικό και σε τεχνικό επίπεδο. Όσον αφορά την Τουρκία και την δήλωση θα ήθελα να πω δύο λόγια για το θέμα αυτό. Η δήλωση αυτή έχει αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα σώζει ζωέ στο Αιγαίο και δεύτερον μειώνει τι μεταναστευτικέ ροέ. Ζητάμε από την Τουρκία να εντείνει τις ε, προσπάθειές τους όσον αφορά τις ε, νέες διαδρομές που εμφανίζονται στην Κύπρο. Πάνω από 24.000 ε, Σύριοι πρόσφυγε που χρειάζονται προστασία έχουν εγκατασταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την δήλωση. Η Κομισιόν τακτικά ζητά από την Κομισιόν να εφαρμόσει τη Συμφωνία Επανεισδοχή πλήρω. και προ όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα ε, έχει τη σημασία του και στον διάλογο για την απελευθέρωση τη ΒΙΖΑ. Όσον αφορά τώρα τι επιστροφέ στην Τουρκία, πρέπει να επιταχυνθεί ο ρυθμός τους. Μέχρι στιγμής έχουν επιστραφεί γύρω στα 360 άτομα από τα νησιά στην Τουρκία. Συνολικά 2.500 άτομα από τον Μάρτιο του 2016. Οι αρχές ε, της Ελλάδας ε, δίνουν προτεραιότητα στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. Σχεδόν 11.500 άτομα έχουν επιστραφεί σε τρίτες χώρες από τον Μάρτιο του 2016 μέσω και των εθελοντικών επιστροφών που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και προγραμμάτων επανένταξης. Τώρα, για το μέσο για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή φιλοξενεί, όπως όλοι ξέρετε, πάνω από 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. 3,6 από τους οποίους είναι Σύριοι. Και καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να τους δώσει ανθρωπιστική βοήθεια και αναπτυξιακή βοήθεια η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μέσω του σχετικού μέσου είναι βασικό κομμάτι της συνεργασίας μας με την ε, χώρα αυτή. Δεν είναι στήριξη την οποία διαχειρίζεται το τουρκικό κράτος, αλλά διαχειρίζονται οι διεθνείς εταίροι μας επί που για τα 4 εκατομμυρία ανθρώπους αυτούς με πολύ απτά αποτελέσματα. Η χρηματοδότηση αυτή συνεισφέρει στην βελτίωση των συνθήκων ζωής και στην προστασία των Σύριων προσφύγων και των κοινοτήτων που τους φιλοξενούν στην Τουρκία. Παραδείγματο χάρη, έχει παρασχεθεί πρόσβαση στην εκπαίδευση για εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά και πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες έχουν λάβει βοήθεια σε ρευστό για τις καθημερινές τους ανάγκες. στήριξή μας Επίσης έχει βοηθήσει στην οικοδόμηση εγκαταστάσεων και στη χρηματοδότηση υπηρεσιών υγείας. Κάνατε ένα σημαντικό ερώτημα για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η πλειοψηφία της χρηματοδότησης ε, γίνεται βεβαίω μέσω κοινή διαχείρισης με τα κρατη Τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να ωφεληθούν από την χρηματοδότηση αυτή που διαχειρίζεται άμεσα η Κομισιόν. Αυτή τη στιγμή υποστηρίζουμε τοπικές και περιφερειακές ε, κοινότητες. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση όπου έχουμε κοινότητες ή περιφέρειες οι οποίες μπορούν να λάβουν μέρος σε έργα ως συνδικαιούχοι. Επίσης, μεγάλο κομμάτι της χρηματοδότησης έχει άμεσο αντίκτυπο σε περιφέρειες ε, και κοινότητες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η διαχείριση του Καρατεπέ, την είπατε του ΙΕ Λέσβο και ο γενικός ε, συντονισμός και η χρηματοδότηση προς την Λέσβο. Και μετά η επέκταση των συστημάτων ίδρυυσης στο βαθύ της ΣΑΜ για να ανακαλύψει τις ανάγκες και της πρωτεύουσας της νήσου και του hotspot. Και μετά υπάρχει το έργο στην Ιταλία που στόχο έχει να καταπολεμηθεί η εκμετάλλευση των μεταναστών στην μαύρη εργασία. Η πρόταση, λοιπόν, για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης για την περίοδο 2021-2027 περιλαμβάνει διατάξεις για την ενίσχυση της εμπλοκής των τοπικών αρχών στον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό των προγραμμάτων. Επίσης ε, περιλαμβάνει κίνητρα για τα κράτη-μέλη όπως υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης σε προγράμματα ένταξης που εφαρμόζουν τοπικές αρχές ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Όσον αφορά τώρα την ε, ανάκτηση των 27.000 ε, θα την καταβάλει η Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα. Οι υπηρεσίε μου θα προετοιμάσουν έναν κατάλογο όλων των άλλων, λίγων είναι, διαταγών ανάκτησης που εκκρεμούν. Όσον αφορά τώρα τον έλεγχο της Κομισιόν, οι έξι αποκεντρωμένες υπηρεσίες για τις οποίες είναι υπεύθυνη η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών έχουν δική τους νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το καταστατικό τους και διοικούνται από ένα ΔΣ που αποτελείται από τα κράτη-μέλη και δύο εκπροσώπους της Κομισιόν. Η Κομισιόν δεν μπορεί να ασκήσει βέτο σε αποφάσεις που λαμβάνουν τα διοικητικά συμβούλια για την παρακολούθηση του έργου των υπηρεσιών αυτών. Η Κομισιόν έχει αναπτύξει μια στρατηγική έλεγχου που αφορά ακριβώς την παρακολούθηση των υπηρεσιών αυτών που λαμβάνουν λεφτά από τον κοινωτικό προπολογισμό. Οι υπηρεσίες ε, έχουν κάθε μία την δική της απαλλαγή για την εφαρμογή του προπολογισμού τους. Για τον σκοπό αυτό Υπάρχει μια ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, ε, την οποία εγκρίνουν τα ΔΣ και αποστέλλεται κάθε χρόνο σε Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Είναι η βάση για την απαλλαγή. Με ρωτήσατε επίσης για την ε, διακίνηση ανθρώπων. Η ανακοίνωση που ήρθε σε συνέχεια της στρατηγικής 2012-2016 καθορίζει συγκεκριμένες στοχευμένες προτεραιότητες και δράσεις οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν βραχυπρόθεσμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέδειξε περαιτέρω λοιπόν ότι δεσμεύεται για την καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων και θεωρεί ότι είναι μεταξύ των προτεραιότητων και των δράσεών τους μέσω της εντολής ε, του συντονιστή καταπολέμησης της διακίνησης που συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη, την κοινωνία των πολιτών και διεθνείς οργανώσεις και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Τώρα, όσον αφορά προγράμματα που έχουμε σε εξέλιξη με τη Γενική Διεύθυνση Home, ε, χρηματοδότηση 4,68 εκατομμύριων για την καταπολέμηση των εγκλημάτων και την βοήθεια στα θύματα. Επίσης, στατιστικά και έκθεση Προέδρου για το 2018 και κατευθυντήρες γραμμές προσφάτως για προστασία των παιδιών και ε, ε, εποπτεία της Ευρωπαϊκής Δράσης 2017-2018, η οποία δημοσιεύθηκε προστάτως. Και να σας πω και δύο λόγια για την επανεγκατάσταση. «34.700 μετανάστες επανεγκαταστάθηκαν από το 2015». 12.700 από την Ιταλία και 22.000 από την Ελλάδα. Πέρσι είχαμε 1.506 άτομα ε, από την Ιταλία και την Ελλάδα βάσει των αποφάσεων ε, του 2015. Περίπου το 95% των ε, επιλέξιμων ετούντων μετεγκαταστάθηκαν με επιτυχία. Είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε περαιτέρω εθελοντική μετεγκατάσταση μέσω χρηματοδότησης. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε σε μέτρα ad hoc και οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στη μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος ευρωπαϊκού ασύλου, ε, μια συνολική δέσμη μέτρων που βασίζεται στην αρχή της ελληνική και του επιμερισμού των ευθυνών. Τώρα, όσον αφορά την επανεγκατάσταση, υπάρχει ένα νέο ε, σύστημα το οποίο ξεκίνησε το 2017. Έχουμε λάβει πάνω από 50.000 τίματα, από, δεσμεύσεις συγγνώμη, από 20 κράτη-μέλη το 2018 και το 2019. Από τις 7 Οκτωβρίου του 2019, 39.000 παρακαταστάσεις είχαν γίνει ήδη βάσει του προγράμματος και έτσι έχουμε ποσοστό εφαρμογής περίπου 78%. Είναι διαθέσιμα 500 εκατομμύρια από ευρωπαϊκά κονδύλια για να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη για τις προσπάθειες επανεκατάστασης και παρά τα καλά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέσω των ad hoc ρυθμίσεων, χρειάζεται ένα διαρθρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανεγκατάσταση. Όσον αφορά τα hot spots στην Ιταλία, θα ήθελα να πω δύο λόγια μετά από την περαιτέρω μείωση των αφήξεων το 2018 και το 2019, το σύστημα υποδοχής πρώτης γραμμής της Ιταλίας ε, δέχτηκε πολύ λιγότερες πιέσεις από ό,τι το 2017. Συνήθως ε, μένουν μετανάστες που περιμένουν μόνο για θελοντική επανεγκατάσταση στα hot spot και θα διοργανωθεί και ένα τεχνικό γύρο τραπόζη στην Ιταλία ε, για να κάνει ένα απολογισμό της παρούσα κατάστασης και να δούμε πιθανά μέτρα για καλύτερη διαχείριση νέων αφήξεων. σχεδόν ολοκλήρωσαμε τις απαντήσεις. Ε, είχαμε πάρα πολλές και διάφορες ερωτήσεις, αλλά ήταν όλες πάρα πολύ σημαντικές, πιστέψτε με. Ελπίζω ότι δεν ξεχνάω κάποιες. Όσον αφορά τα χαμηλά ποσοστά απορρόφηση σε κάποια κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει την υποστήριξή της συνεχώς, προκειμένου να βελτιώσουμε τα ποσοστά εφαρμογής, ιδίως ε, για τις πιο κατεπίγουσες ε, περιπτώσεις. Αναφερθήκατε επίσης ε, σε μετανάστες στη Λιβύη και την κατάσταση στη Λιβύη. Εδώ μπορώ να σας πω ότι η κατάσταση εξακολουθεί να είναι χαόδης και δύσκολη σε πολιτικό επίπεδο. Και χάρη στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από το ε, κατεπήγον καταπίστευμα για τη Βόρεια Αφρική και ε, χάρη και στη δράση των Ηνωμένων Εθνών είχαμε τα εξής αποτελέσματα ξεκίνησε να λειτουργεί εγκατάσταση ε, συγκέντρωσης και αναχώρησης ε, στην ε, Τρίπολη. υπάρχει ένα σύστημα για τη διεθνή προστασία και ένα σύστημα διεθνών επιστροφών πάνω από 40.000 μεταναστών από το 2017. Η πολύ σημαντική δουλειά που κάνει η Λιβική ακτοφυλακή διασώζει ζωές και είχαμε πάνω από 800 άτομα το 2019. Και τέλος, Όσον αφορά το ποσοστό των επιστροφών, το 2018 το ποσοστό επιστροφών μειώθηκε στο 63% σε σχέση με το 36,79% που είχαμε το 2017. Είναι σαφές ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτή η μείωση είναι εύκολο να εξηγηθεί ε, λόγω του χαμηλότερου αριθμού των υπηκών τρίτων χωρών που ε, ε, παραμένουν λιγότερο και έτσι έχουμε μικρότερο ποσοστό επιστροφών στις χώρες αυτές περιπτώσεις αυτές ήταν πάνω από το 100% στις προηγούμενες χρονιές, γι' αυτό και είχαμε αύξηση των ποσοστών. Τα έχουμε απαντήσει όλα αυτά και στις ερωτήσεις ε, για την απαλλαγή από το ελεκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. ο κύριο Μπρίνκχαρτ ε, τώρα. Θέλετε κι εσείς να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Κατάλαβα ότι υπήρξε μία μόνο ερώτηση που αφορούσε άμεσα το ε, ελεγκτικό συνέδριο. Κατά τη γνώμη μας, οι εθνικές αρχές έχουν διαφορετικά επίπεδα αρμοδιοτήτων ανάλογα με το πώς ε, είναι δομημένες οι αρμόδιες αρχές και πώς είναι στελεχωμένες επίσης. Έχουμε ελέγξει τα συστήματα και την τεχνική αρρωγή σε 8 κράτη-μέλη και για να είμαστε δίκαιοι δεν βρήκαμε σημαντικά προβλήματα. Βρήκαμε ότι χρειάζονται βελτιώσεις στη διαχείριση των συστημάτων των κρατών μελών και έχουμε περιλάβει συγκεκριμένες ένδειξεις ε, ε, και υποδείξεις ε, στις εκθέσεις μας. Μετά από μια αργή αρχή τα κράτη-μέλη προχωρούν πιο γρήγορα και όχι με την ταχύτητα που θα επιθυμούσαμε. Τα ποσοστά τα, ε, ε, βέβαια εκτέλεσης μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω. Για την απλοποίηση καλωσορίζουμε την πρόταση για ένταξη του MVISF στην ε, κανονισμό κοινών διατάξεων και βέβαια καλωσορίζουμε τα νέα μέτρα που προτείνονται για το νέο πολιετές πλαίσιο. Σας ευχαριστώ. Έχουμε κάποιους ακόμα που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Χριστοφόρου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακούοντας τις ολοκληρωμένες απαντήσεις που έδωσε προλίγου ο Επίτροπος για το Migration, ο κύριος Αβραμόπουλος, πέρασαν από το μυαλό μου και από μπροστά μου οι τραγικές και ανεξέλεκτες εικόνες με το προσφυγικό πριν πέντε χρόνια όταν ήταν μόλις αναλάβανε τα καθήκοντα του Επιτρόπου. Για να μπορέσουμε πραγματικά να αποτυπώσουμε και το έργο που επιτελέστηκε αλλά και την προσπάθεια του κάθε Επιτρόπου πρέπει να δούμε τι επαραλάβανε πριν ακριβώς πέντε χρόνια. Χωρίς σχέδιο, ξέφραγον να μπαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πάντες των υποπανικών είχε ενώπιον του να διαχειριστεί όχι μόνο τους πρόσφυγες που έρχονταν κατά κύματα και δυστυχώς δημιουργούνταν εκείνες οι τραγικές συνθήκες και καταστάσεις, αλλά είχε ενώπιον του να αντιμετωπίσει την Τουρκία, μια Τουρκία η οποία ουδέποτε ευαισθητοποιήθηκε για το προσφυγικό, για το προσφυγικό, αλλά χρησιμοποιήσαμε σήμερα το προσφυγικό αυτόν το ανθρωπιστικό θέμα για να το εκμεταλλευτεί, για να εφαρμόσει τι πολιτικέ και τι στρατηγικέ τη. Και έχει απέναντι του Επίτροπο, ο κύριο Αβραμόπουλο, να αντιμετωπίσει αυτήν την Τουρκία, η οποία δεν συνδιαλέγεται, δεν συνομιλεί πολλέ φορέ και δεν αποδέχεται τι αρχέ και τι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την διαχείριση του προσφυγικού που μέχρι σήμερα εκβιάζει για αυτό το ανθρωπιστικό θέμα. Ενώπιον αυτή τη καταστάσεω, θεωρώ ότι υπήρξε η επιβεβλημένη διαχείριση εκείνη για να μην προκληθεί το χάος και να μην υπάρξουν ανεξέλεκτες καταστάσεις. Πέραν αυτό, και όλοι μας θα πολλές φορές προς την Επιτροπή τι έπραξε περισσότερο για να μην έχουμε τα προβλήματα γιατί τίποτα δεν είναι τέλειο, φυσικά και όλοι εμείς πρέπει να αναρωτηθούμε τι πράξαμε και τι έπραξαν οι χώρες μας για να βοηθήσουν το προσφυγικό και να μην είναι υπόθεση μόνο της Επιτροπής και κάποιων χωρών που έτυχε να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή απέναντι από τις σειράξεις και τους πολέμους στη Μεσόγειο. Τελειώνοντας θα πω ότι θεωρώ ευτύχημα που σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που το προσφυγό είναι το μείζο θέμα και κλείθει η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη της να το αντιμετωπίσει, οι άλλες χώρες που το δημιούργησαν όπως η Ρωσία, η Αμερική και άλλες χώρες, όχι μόνο δεν υποδέχτηκαν ούτε έναν πρόσφυγα, αλλά απαλλάχθηκαν των ευθυνών τους. Θεωρώ ευτύχημα γιατί σε αυτήν την κρίσιμη, στο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο βρέθηκε ο Δημήτρης ο και ως Ευρωπαίοι καμιά φορά πρέπει να αισθανόμεθα περήφανοι όταν τέτοιοι άνθρωποι διαχειρίζονται αυτά τα κρίσιμα ζητήματα και θεωρώ ότι παρά τα λάθη και τις παραλήψεις που μπορεί να έγιναν γενικά από τις χώρες, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορώ να διανοηθώ τι θα επικρατούσε εάν δεν με αποφασιστικότητα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εργαζόμενος νυχθημερών ευρισκόμενο στα παράλια τη Ανατολική Μεσογείου αλλά και στην Τουρκία ταυτόχρονα και όπου χρειαζόταν, δεν έδινε τη μάχη για να υπάρξει αυτή η βελτίωση που υπήρξε μέσα στα πέντε χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον δεν μπορεί να μιλά για ξέφραγο να μπέλει, δημιουργήσε σύνοροφυλακή. Υπήρξαν συμφωνίε, υπήρξε διαχείριση. Και ήθελα να ξέρω και εν είδη ερωτήσεω, εάν σήμερα μέσα από τι νέε συνθήκε και τα νέα δεδομένα η νέα κυβέρνηση τη Ελλάδα με τις νέες αποφάσεις που έλαβε θα υπάρξει καλύτερη διαχείριση του προσφυγικού. Τελειώνοντας θα ήθελα να ερπίζω και είναι πραγματικά ευχή ο νέος Επίτροπος για τα θέματα του migration να διαχειριστεί την όλη κατάσταση με την αποφασιστικότητα, την δεξιοτεχνία, την πραγματικά νυχθημερή προσπάθεια του Επιτρόπου και των συνεργατών του που μπορεί να μην είχαμε το τέλειο αποτέλεσμα, αλλά μη τι άλλο δεν θυμίζουμε τις μέρες πριν πέντε χρόνια όταν αναλάβανε ο σημερινός Επίτροπος. Και θα ήθελα να ξέρω και ποια είναι η άποψή του όσον και αν δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις για αυτά τα ζητήματα, για την περαιτέρω διαχείριση του ζητήματος, για τυχόν επιδείνωση ή για τυχόν βελτίωση, γνωρίζοντας όλα τα δεδομένα και με την Τουρκία αλλά και με τη διαχείριση που τη χάνει από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Muchas gracias. Σας ευχαριστώ πολύ. El señor Adinolfi. Ο κύριος Αντινόλφη. Grazie. E, ho ascoltato le parole del commissario. Άκουσα τα λόγια του Επιτρόπου. Όμως από τα στοιχεία που έχω λάβει από την ΥΠΑ Τερμοστία του ΟΗΕ για το 2018, λένε λοιπόν αυτά τα στοιχεία ότι τους πρώτους έξι μήνες του 2018 είχαμε 13.000 600 μετανάστες και στην Ελλάδα 12.000. Αυτά τα στοιχεία έχει η πατερμοστία για τους πρόσφυγες του ΟΗΕ. Αν λοιπόν συγκρίνουμε τα νούμερα που δόθηκαν στην Ελλάδα 2 δις 2 ενώ 1 δις μόνο δόθηκε στην Ιταλία το 2018 αν τα συγκρίνουμε αυτά τα στοιχεία να πω ότι δεν αντιστοιχούν στους μετανάστες που έχουν φτάσει. Θέλω να ξέρω λοιπόν Πώς γίνεται να έχουμε τέτοια διαφορά ανάμεσα στα χρήματα που δόθηκαν στην Ελλάδα και τα νούμερα που δόθηκαν στην Ιταλία και που όπως είπα τα βασίζω στα ε, νούμερα που πήρα από την ύποτη αρμοστία για τους πρόσφυγες του ΙΕ. Το ίδιο και για τους μετανάστες που μειώθηκαν στην Ιταλία. Ίσως οι Ιταλικές πολιτικές που ασκήθηκαν από την Ιταλική κυβέρνηση από το Μάρτιο του 2018 μέχρι τον Ιούλιο του 2019 να οδήγησαν στη μείωση της μετανάστευσης. Τώρα, όσον αφορά τα ασφάλεια και δηλαδή τα εγκλήματα στο ψηφιακό κόσμο, είναι ένα πρόβλημα εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο αφορά όλες τις εταιρείες και όλους τους ιδιώτες, αλλά και τα ίδια τα κράτη. Εάν τα χρήματα που χορηγήθηκαν από τον προπολογισμό το 2018 αρκούν για να αντιμετωπιστούν τα ψηφιακά ε, αδικήματα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κινίτσι. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους φιλοξενούμενους μας και κυρίως τον Επίτροπο Αβραμόπουλο για την εργασία του στο θέμα της μετανάστευσης και με ιδιαίτερη αναφορά στους ε, συνόδευτους ε, ανήλικους. Είναι ένα θέμα το οποίο επεξεργάστηκε με θεσμική ευαισθησία αλλά και προσωπική ευαισθησία και να τον ευχαριστήσω για τη χώρα μου, την Ιταλία, όπου η δέσμευση για υποδοχή, στήριξη και ένταξη των ανηλίκων ήταν ε, ε, σημαντική και νομίζω πως έφερε καλά αποτελέσματα τα μέτρα τα οποία υιοθετήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμα και αν βέβαια δεν ήταν ε, πλήρη και εξαντλητικά, μας επέτρεψαν να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα για το οποίο έχουμε επανειλημμένα συζητήσει και επί το οποίο βρήκαμε ευαισθησία αυτό που αφορά δηλαδή τους εξαφανισμένους ανήλικους, ε, δηλαδή αυτούς για τους οποίους έχουν χαθεί τα ίχνη από τη στιγμή που έχουν έρθει στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Όμως σας ρωτώ, θεωρείτε πως υπάρχουν ακόμα μέτρα προτεραιότητας που μπορούμε να λάβουμε σε σχέση με τους ανήλικους και ε, σε σχέση με τη διακίνηση ανθρώπων. Ξέρουμε πως οι ανήλικοι είναι τα πιο ευάλωτα θύματα και αυτά τα οποία τραυματίζονται και περισσότερο λόγω της εμπορίας ανθρώπων. Είναι ένα δραματικό φαινόμενο. Σας ρωτώ υπό το φως της εμπειρίας σας και με βάση τις εργασίες που έχετε κάνει πώς είναι δυνατόν να βελτιώσουμε την προστασία των ανήλικων μεταναστών, ποια μέτρα θα πρέπει πρέπει ακόμα να λάβει η Επιτροπή, ώστε να παρέχει την κατάλληλη προστασία στους ανήλικους που φεύγουν με δραματικές καταστάσεις, από μάλλον δραματικές καταστάσεις. Ε, πώς μπορούμε λοιπόν εμείς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τους υποδεχτούμε και να τους εντάξουμε στις χώρες μας. Ευχαριστώ. Muchas gracias. De σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω και πάλι λοιπόν το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει σε αυτές τις ε, ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω απαντώντας στον κύριο Χριστοφόρου στα ελληνικά. Κύριε Χριστοφόρου, είναι σωστό αυτό που είπατε και θυμήσατε πώς ξεκινήσαμε πριν από πέντε χρόνια. Είσαστε και εσείς εκεί και από τη δική σας σκοπιά δίνατε καθημερινά τη μάχη για να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία ευνηδίασε την Ευρώπη. Και θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ούτε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, αλλά ούτε και τα κράτη-μέλη μπορούσαν να ανταποκριθούν εκείνη την ώρα όταν ευνηδιάστηκαν από αυτές τις αθρώες αφήξεις κοντά ενός εκατομμυρίου ανθρώπων που πέρναγαν είτε από τον αποκαλούμενο κεντρικό ευρωπαϊκό ε, μεσογειακό διάδρομο ή από το Αιγαίο. Τότε ήταν που η Επιτροπή, η οποία πρέπει να σας πω δεν είχε στρατηγική για την μετανάστευση, αλλά ούτε και για την ασφάλεια, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα υιοθέτησε με την βοήθεια κυρίως πρέπει να το πω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν από το ξεκίνημα ο ισχυρότερος σύμμαχός μας, την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια και τη Μετανάστευση. Ήρθαν λοιπόν τα γεγονότα, όπως αργότερα και τα δραματικά γεγονότα, πέντε μήνες μετά, με τις τρομοκρατικές ενέργειες. Τα καταφέραμε όμως. Και θέλω να πιστεύω ότι αφήνει αυτή η Επιτροπή μια πολύ ισχυρή κληρονομιά για την επόμενη διότι όλα αυτά που συντελέστηκαν και που δεν είναι τη στιγμή να τα παριθμίσω, είναι αυτά που έδωσαν απάντηση στις μεγάλες προκλήσεις. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες, θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό όμως. Πώς θα ήσαν τα πράγματα και ποιες θα ήσαν οι εξελίξεις αν δεν είχαν αναλυθεί όλες αυτές οι πολιτικές πρωτοβουλίες. Μια παρατήρηση μόνο πολιτικής αξίας θέλω να κάνω. Τελικά, δεν ήταν η οικονομική κρίση που έφεται σε αμφισβήτηση το ευρωπαϊκό σχέδιο, το European Project, αλλά περισσότερο η προσφυγική κρίση και η κρίση ασφάλειας. Διότι δοκιμάζονταν ευθέως οι αρχές και οι αξίες πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε το ευρωπαϊκό, η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική τα τελευταία 60 χρόνια. Οι αρχές της αλληλεγγύης, και της ευθύνης, της υπευθυνότητας. Ήταν λοιπόν πολύ δύσκολο, αλλά επαναλαμβάνω ότι καταφέραμε πολλά, χωρίς να σημαίνει ότι το πρόβλημα λύθηκε, διότι δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει, κύριε Χριστοφόρου, το μέλλον. Η γεωπολιτική αστάθεια είναι ακόμα εκεί και οι βασικές αιτίες που προκάλεσαν τα προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα είναι ακόμα εκεί και η ευθύνη είναι συλλογικά του κόσμου ολόκληρου. Στην αρχή όλοι πίστευαν ότι είναι ένα ζήτημα του Ευρωπαϊκού Νότου. Ένα πρόβλημα τη Ιταλία, τη Ελλάδα, τη Μάλτα και τη Ισπανία. Πολύ σύντομα καταλάβανε όλοι ότι είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα που απαιτούσε ευρωπαϊκέ λύσει, αλλά και ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα με παγκόσμιε διαστάσει. Την ώρα που είμαστε εμεί εδώ, αξίζει να γνωρίζετε ότι κοντά 400 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο είναι σε κίνηση. They are on the move. Είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι μετανάστες. Και αυτό θα είναι ένα ζήτημα που θα απασχολήσει την παγκόσμια κοινότητα και γι' αυτό είχαμε πάρει την πρωτοβουλία πριν από τρία χρόνια να ζητήσουμε εγώ προσωπικά από τον τότε Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να συγκαλέσει μια παγκόσμια διάσκεψη, μια έκτακτη γενική συνάντηση του ΟΗΕ, κάτι το οποίο και έγινε. Το ίδιο και για την ασφάλεια, όπου έπρεπε πολλά να γίνουν, διότι όπως είπα και στα εισαγωγικά μου, μπορεί να ιτήθηκε η τρομοκρατία επί του εδάφους, αλλά δεν έχει ιτηθεί ακόμα στο νέο πεδίο μάχης που είναι το ίντερνετ. Ιδρύσαμε λοιπόν, ήταν μια πρωτοβουλία που πήρα το Internet Forum, το οποίο έφερε κοντά σε μια σχέση αγαστής συνεργασίας και σχέση εμπιστοσύνης τους βασικούς Internet providers, τις μεγάλες πλατφόρμες του ίντερνετ, Facebook, Twitter, ε, Microsoft και τις άλλες, σε μια συνεργασία που έχει αποτελέσματα. Το τρομοκρατικό υλικό που οδηγεί στη ριζοσπαστικοποίηση κατεβαίνει πλέον από τις μεγάλες πλατφόρμες μόλις εμφανιστεί μέσα σε μία ώρα. Εξαιρετική συνεργασία. Αυτός ο αγώνας, αυτή η προσπάθεια όμως πρέπει να συνεχιστεί, διότι η απειλή της τρομοκρατίας υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν ασφάλεια και πρέπει να την έχουν και αυτή είναι μία από τις βασικές αποστολές που έχουν αναλάβει τα ευρωπαϊκά όργανα με πρώτη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως είπαμε αρρωγό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια παρατήρηση όμως επίσης πολιτική πρέπει να αντιληφθούν τα κράτη-μέλη ότι έχουν τεράστιες ευθύνες. Η κριτική που ασκείται κατά καιρού είναι εναντίον της Ευρώπης. Αόριστα. Αλλά η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο έχει εδώ του εκπροσώπους της. Και πρέπει να πω ότι οι εκπρόσωποι όλων των πολιτικών παρατάξεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάνουν εξαιρετική δουλειά και είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι. Αλλά οι κυβερνήσει καμιά φορά δεν συμφωνούν κάνω μια διάκριση ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τι κυβερνήσει του. Γιατί οι κυβερνήσει έρχονται και απέρχονται. Τα κράτη όμω μένουν. και να καταλάβουν ότι έχουν μεγάλη ευθύνη να κρατήσουν όρθια την Ευρώπη. Κυρίω στην αντιμετώπιση αυτών των τόσο σημαντικών ζητημάτων. Για την ελληνική κυβέρνηση, ο τελευταίο νόμο που πέρασε είναι στη σωστή κατεύθυνση. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αρχίσει να δίνει αποτελέσματα. Έχουν πλήρη επίγνωση της καταστάσεως και εμείς θα συνεχίσουμε να βοηθούμε όχι μονάχα τις ελληνικές αρχές αλλά και τις αρχές όλων των χωρών που είναι κάτω από πίεση. And now I go, I turn again to English. I would like to refer to the support of uh, Cyprus. Cyprus is on the top of our priorities because Cyprus η Κύπρος, η Κύπρος είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Έχουμε λάβει μέτρα ώστε να επιτείνουμε οικονομικά ε, την ε, βοήθεια προς την Κύπρο και την επιχειρησιακή βοήθεια. 91 εκατομμύρια ευρώ ε, καθώς και 12 εκατομμύρια για δυνατότητες υποδοχής και άλλες δραστηριότητες σχετικέ με το άσυλο. Στα τέλη του 2018 η Κομισιόν έδωσε ακόμα 3,1 εκατομμύρια ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητα υποδοχής. Εν ώψη νέων μεταναστευτικών ροών, η Επιτροπή θα είναι έτοιμη να εξετάσει έτοιμα για περαιτέρω χρηματοδότηση υπό την επίγουσα ε, βοήθεια. Η Κύπρος, η κύριε Χριστοφόρου, θα λάβει μέσα στο 2019 επιπλέον στήριξη υπό το πρόγραμμα εσωτερικής ασφάλειας, ώστε να ε, βελτιώσει το ΣΥΣ και να αναπτύξει διάφορα συστήματα ε, ίντερνετ μαζί με τους οργανισμούς, την ΕΑΖΟ, την Europol, την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή θα συνεχίσουμε και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε περισσότερα αν χρειαστεί. Επίσης είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την εφαρμογή ε, ε, θελοντικών προγραμμάτων ε, τη βάση διμερών συμφωνιών. Κύριε Αντινόλφη, τα νούμερα δεν είναι τα ίδια, σίγουρα. Η Κύπρος, η Ιταλία και η Ελλάδα και οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος δεν είναι, και δεν, δεν είναι μόνα και δεν θα φεθούν μόνα. Έχουμε διαρκώς προσφέρει οικονομική, τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια με ειδικού που μεταβαίνουν επί τόπου και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε θα συνεχίσουμε δεν να χρηματοδοτούμε την εθελοντική μεταγκατάσταση. Γι' αυτό και η πολιτική μας προτεραιότητα είναι η δημιουργία ενός δικαιού και αποτελεσματικού συστήματος ε, ασύλου. Για την Ιταλία, θα σας πω ότι από την πρώτη μέρα ήμουν και παραμένω σε στενή συνεργασία με τις Ιταλικές κυβερνήσεις. Έχω συνεργαστεί πολύ καλά και πολύ αποτελεσματικά με τον Υπουργό Μινίτη και με, βεβαίως με τον Υπουργό ε, Σαλβίνη και ε, στην αρχή με τον κύριο Αλφάνη. Η Ιταλία θα πρέπει να είναι περήφανη γιατί έχει δείξει δέσμευση και έχει ε, δράσει πολύ πολύ αποτελεσματικά και θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον Ιταλικό λαό. Μαζί με τον ελληνικό λαό έχουμε δείξει τι σημαίνει όταν λέμε ανθρωπιά και ευθύνη στην Ευρώπη. Οι λαοί των δύο αυτών χωρών θα πρέπει να επενεθούν για τον τρόπο με τον οποίο φέρθηκαν τα χρόνια αυτά. Κυρία Κινίτσι. Να σας πω κάτι πολύ απλό. Αυτά που είπατε τα λέω τα τελευταία πέντε χρόνια, όχι εδώ μόνο, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και τα λέτε και εσείς. Και θέλω θερμά, θερμά να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική προσωπική σας δέσμευση, ιδιαίτερα για τους ανηλίκους. Δεν διστάζω να σας πω ότι ήσασταν εκείνοι που με ευαισθητοποιήσατε εξ αρχής, όταν προσπαθούσα να ε, καταλάβω τι πρέπει να κάνω και πώς ήσασταν εσείς πρωτοπόρος και νομίζω πως το Κοινοβούλιο και η Ευρώπη σας χρωστάν πολλά ε, σε εσά προσωπικά. Χαίρομαι που ε, είστε και πάλι στο Ευρωκοινοβούλιο και είμαι βέβαιος ότι θα παίξετε πολύ σημαντικό ρόλο και για το μέλλον. Αναφερθήκατε στη κατάσταση των ανελίκων στην Ελλάδα. Ε, η ασφάλεια, όπως είπα, και η προστασία των ανηλίκων, ιδιαίτερα των ασυνόδευτων ανηλίκων, θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα για όλους μας. Το λέμε αυτό και το επαναλαμβάνουμε. Το λέμε και το επαναλαμβάνουμε σε με όλες τις αρχές των κρατών μελών. Πρέπει να αναλάβουμε δράση και η κατάσταση αυτή ε, είναι γνωστή σε όλα τα κράτη-μέλη. Το αναφέρουμε διαρκώς σε πολυάριθμες εκθέσεις. Μια από τις προτεραιότητες ε, του, της ε, έκλεισε για υποβολή προτάσεων είναι, για, ήταν για να ε, γίνουν διάφορες διακρατικές δράσεις και ε, η μία εξ αυτών ήταν για τους ε, ανήλικους και κυρίως τους ανισυνόδευτους ανήλικους. Θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα το 1η Δεκεμβρίου. Επίσης υπάρχει ακόμα μία ε, ένας διαγωνισμός για τα παιδιά και την προστασία τους. Κυρία Κινίτση, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση για αυτό το ζήτημα με τον τρόπο που το κάνετε εσείς, γιατί πρόκειται για παιδιά, πρόκειται για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και πριν να κλείσουμε... Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα, κυρία Ούνιφιλ, ο, τελική σας παρατήρηση. Señora Winzig, no me escucha. Señora Winzig, ¿quiere decir algo para finalizar? No. Θέλετε να πείτε κάτι για να κλείσετε τη συζήτηση, όχι. Ωραία. Λοιπόν, Κύριε Επίτροπε, μάλλον θα είναι η τελευταία σας ε, παρέμβαση στην Επιτροπή μας και γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά σας, τη συμβολή σας και την προσήλωσή σας στις ευρωπαϊκές αξίες. Να σας ευχαριστήσω επίσης για την αγαστή συνεργασία που είχαμε ανέκαθεν εδώ και να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Να ευχαριστήσω επίσης όλα τα μέλη της Επιτροπής, τον κύριο Μπρίνχαρτ ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου για αυτή την πολύ ζωντανή και ε, πλούσια συζήτηση και να πω ότι θα λάβουμε υπόψη αυτό το σχέδιο έκθεσης και θα το εξετάσουμε στις 20-21 Ιανουαρίου του 2020. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο. Vamos a hacer un breve receso de unos minutos. περάσουμε στο επόμενο σημείο, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα ολίγων λεπτών. Continuamos la sesión. Συνεχίσουμε. Τώρα έχουμε την ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Χάν, που είναι αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική. Ε, με χαρά σας καλωσορίζουμε κύριε Χάν. Ο κύριος Χάν υπέβαλε ε, μάλλον συγγνώμη, ανέλαβε αυτή την επιπλέον εργασία ως Επίτροπος ε, για την Περιφερειακή Πολιτική, γιατί η κυρία Κρέτου εξελέγει εδώ Ευρωβουλευτής. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για τη διαθεσιμότητά σας, για την ευελιξία σας να έρθετε σήμερα εδώ. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, οι απαντήσει στο ερωτηματολόγιο που σας στείλαμε εκ των προτέρων έχουν διανεμηθεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής μας και σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω τον κύριο κύριο Μέρφυ που είναι μέλος ε, του ελεγκτικού συνεδρίου και ταυτόχρονα του δίνω το λόγο ώστε να μας πει ποιες είναι οι εντυπώσεις του για περίπου 10 λεπτά. Κύριε Μέρφυ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, με χαρά βρίσκω αυτή την ε, νέα καινούργια επιτροπή του Ευρωπαϊκού για, θα σας μιλήσω για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική σύγκληση με βάση τη διαχείριση της DG Regio και επασχόληση σύμφωνα με το νέο ελεγκτικό πλαίσιο για την περίοδο 2020 και για να γίνει μεγαλύτερη χρήση των πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά και να μειωθεί το διοικητικό, ο διοικητικός φόρτος στους τελικούς δικαιούχους, διατηρήσαμε την ίδια προσέγγιση για το 2018 όπως και για το 2017. Αυτό το νέο πλαίσιο ε, προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη και οι αρχές τους επιβεβαιώνουν ότι το υπόλοιπο, το είναι κάτω από το 2% ανά ε, συναλλαγή και ανά επιχείρημα. Ε, και στο τέλος βλέπουμε εμείς αν έχουμε μείνει κάτω από τα ποσοστά αναφοράς. Ο στόχος του ελέγχου ήταν διφυής, να συμβάλλουμε στο πιστοποιητικό ασφάλειας και να αξιολογήσουμε το νέο πλαίσιο για ελέγχους και ασφάλεια και το βαθμό στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό. Γι' αυτό το φετινό, λοιπόν, τη φετινή δήλωση λοιπόν έχουμε εξετάσει ένα δείγμα 220 συναλλαγών εκ των οποίων αφορούσαν την DG ε, Regio. Όλες ε, οι δοκιμές αφορούν άλλους ε, πληθυσμούς τους οποίους καλύπτουν οι δικές μας DG. Τα κράτη-μέλη και οι ελεγκτικές αρχές είχαν προηγουμένως ελέγξει και έχουν αναθεωρήσει τους καταλόγους τους καθώς και τις αποδείξεις που είχαν για να, στις οποίες βάσισαν τα αποτελέσματα του ελέγχου και τις νομοδοτήσεις τους. Εμείς εντοπίσαμε 36 σφάλματα που δεν είχαν ανοιχνευτεί από τις ελεγκτικές αρχές των κρατών. Λαμβάνοντας υπόψη τα 60 σφάλματα που βρήκαν οι ελεγκτικές αρχές των κρατών μελών και τα διόρθωσαν πράγμα που ανήλθε σε 314 εκατομμύριο ευρώ που καλύπταν τις δύο προγραμματικές περιόδους εκτιμούμε το επίπεδο σφάλματος ε, στην υποκατηγορία 1β να είναι 5% σε σύγκριση με το 3% το προερασμένο έτος και 4,8% το προπερασμένο έτος. Γι' αυτό θα ήθελα να θυμίσω ότι το 2017 ήταν μια συνήθιστη χρονιά. Ένα περιορισμένο αριθμό κρατών μελών, δηλαδή 17, είχαν υποβάλει χαμηλό επίπεδο δαπανών και αντιστοιχεία ε, του ERDF και του Ταμείου Συνοχή ε, και οι σχετικέ δαπάνε ήταν πολύ πιο περίπλοκε και χαμηλότερε από ό,τι συνήθω. Φέτο, οι μη επιλέξιμε δαπάνε μαζί με την παραβίαση διαφόρων κανόνων εσωτερική αγορά σε ένα πιο υψηλό επίπεδο σφάλματος. Είναι υψηλότερο λοιπόν και πράγμα το οποίο σημαίνει, συνήθως μάλλον περιλαμβάνει τις διαδικασίες ε, διαγωνισμών, ε, τις ε, υποθέσεις κατοικών ενισχύσεων καθώς και τους εθνικούς κανόνες που παραμένουν περίπλοκοι. Έχουμε λοιπόν διαπιστώσει ότι η Κομισιόν έχει προτείνει 80 μέτρα απλοποίησης μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Εάν ξεκινήσουμε με την αξιολόγηση της εργασίας των 100 μελών, έχουμε να δούμε 126 ελεγκτικά και αρχές και την εργασία μόνο 15 εξ αυτών συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε πως υπάρχει ένα μόνιμο σφάλμα κάτω από το 2% ενώ ορισμένοι είναι πάνω από αυτό το κατόφλι. Μάλιστα 8 από τις 15 που ε, ε, ανάφεραν ε, τα στοιχεία τους έχουν ψηλότερο σφάλμα για την περίοδο 2014-2020. Έχουμε επίσης εντοπίσει προβλήματα και μάλιστα έχουμε διαπιστώσει πως ε, εσφαλμένα έχει αναφερθεί ένα χαμηλό ποσοστό σφάλματος ενώ στην πραγματικότητα είναι πάνω από το 2% το περιθώριο σφάλματος. Επίσης βρήκαμε κάποιες αδυναμίες όσον αφορά τις εθνικές ελεγκτικές αρχές λόγω δειγματοληψίας ε, και έπρεπε να ε, ξανακάνουμε 64 συναλλαγές περιλαμβανομένων 48 σε συγκεκριμένες επιτόπιες ελέγχους. Έχουμε μια κάποια βελτίωση, αλλά χρειάστηκαν επιπλέον πόροι και ε, επιπλέον φόρτος για ορισμένους δικαιούχους. Τα αποτελέσματα των εργασιών της Κομισιόν είναι η βάση δε για την ε, εκτίμηση των σφαλμάτων και για τις ε, επιφυλάξεις που εκφράζονται μέσα στην ετήσια έκθεση. Έχουμε αναθεωρήσει το KPI 5, όπως αυτό αποκαλείται, και αυτό έχει ελεγχθεί με τη νέα ελεγκτική διαδικασία. Έχουμε λοιπόν πιθανές διορθωτικές δράσεις για 40 από τις 175 ε, συναλλαγές που ελέγχονται. Άλλο σημαντικό ποσοστό σφάλματος είναι ο κίνδυνος στην πληρωμή, πράγμα που σχετίζεται με τις δαπάνες συνοχής. Επειδή αυτές οι δαπάνες δεν έχουν υποστεί το νέο κύκλο ελέγχου, η... πρόκειται για προεκβολές οι οποίες ε, θα επαληθευθούν ε, στο μέλλον και δυνητικά θα διορθωθούν. Εν γέννη πάντως, λόγω των μειονεκτημάτων του νέου πλαισίου ελέγχου και ε, πιστοποιητικών ασφαλείας δεν μπορούμε να βασιστούμε στην ετήσια αυτή έκθεση. Έχουμε υποβάλει τρεις συστάσεις για να βελτιώσουμε την κατάσταση στο μέλλον. Τις έχει δεχτεί η Κομισιόν και επίσης αναφερόμαστε σε συστάσεις που κάναμε πέρυσι και αφορούν αυτά τα ίδια ε, προβλήματα. Αγαπητοί κύριοι Ευρωβουλευτέ, είναι σημαντικό να δαπανώνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια σύμφωνα με του κανόνε, αλλά είναι επίση σημαντικό να βλέπουμε αν υπάρχει θετικό αντίκτυπο από τα νέα μέτρα. Ε, στο κεφάλαιο 6 έχουμε εδώ χωριστά εξετάσει τα συστήματα απόδοση ε, των κρατών μελών. Υπάρχουν συστήματα εποπτεία από πλευρά των κρατών μελών, αλλά αρκετέ φορέ οι αρχέ δεν έχουν φτιάξει ε, τους δείκτες με τρόπο ώστε να μετράτε η αποδοτικότητα. Επίσης ξέρουμε πως τα, συμπληρωμένα με, τα ολοκληρωμένα project κάποιες φορές δεν έχουν επιτύχει πλήρως τους στόχους τους. Τέλος, ελπίζουμε πως αυτά τα πορίσματα θα σας είναι χρήσιμα σε σχέση με την συνοχή και το δικαστήριο, να σας πω, πως έχει εκδώσει 13 ειδικέ εκθέσεις και 6 αναθεωρήσεις σε αυτό το τομέα πολιτικής το 2018 και και 19. Η δημοσιευμένη μας νομοδότηση του 2018 δίνει τις απόψεις μας για την προτινόμενη κοινό κανονισμό διατάξεων που διέπει το PDP 2021-2027. Θα ολοκληρώσω τονίζοντας ότι τα σφάλματα που εντοπίζουμε δεν, έχουν, δεν σημαίνουν ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους σωστούς κανόνες και προϋποθέσεις, γιατί τα προγράμματα μπορεί να μην έχουν ακόμα ολοκληρωθεί ή και αν έχουν ολοκληρωθεί να είχαν θετικές επιπτώσεις Πρέπει να τονιστεί πως η απάτη είναι διαφορετική από ένα σφάλμα. Το δικαστήριο αναφέρε νέα υποθέσεις ε, υποψίας για απάτη στην ΟΛΑΦ ε, που μόνο η μία αφορούσε ε, συναλλαγή της συνοχής από το 2017. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Χολμάιρ που δυστυχώς δεν είναι σήμερα εδώ και επίσης να ευχαριστήσω για την συνεργασία στη διάρκεια της ε, διαδικασίας δεν είναι πάντοτε εύκολο γιατί είναι πολύ περίπλοκη αυτή η κατάσταση η, και ο τομέας της πολιτικής και συχνά απαιτείται επαγγελματική κρίση. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον Επίτροπο. Κυρία Χάν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αξιότιμε κύριε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να λάβω το λόγο εδώ σήμερα. Πρέπει να πω ότι νιώθω σαν στο σπίτι μου μετά από πέντε χρόνια, αλλά Με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η αιτιολογημένη γνώμη του ελεκτικού συνεδρίου για το 2018 ήταν ότι το ποσοστό σφαλμάτων οδηγεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλο ένα και πιο κοντά στο ε, κατόφλι. Όπως ε, είπε και το ελεκτικό συνέδριο, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι υποστηρίξαμε την Πρόεδρο για τα επόμενα χρόνια και αυτό περιλαμβάνει και την πολιτική συνοχή που διαδραμάτισε ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Το δικαστήριο αναγνώρισε τι κοινέ μα προσπάθειε και τις ε, καλέ πρακτικέ μα και ε, την ανάγκη για περαιτέρω βελτιώσει. Θα ήθελα να σα αναφέρω τέσσερι βασικέ παρατηρήσει πριν περάσουμε στη συζήτηση. Πρώτον, ε, ποσοστό σφαλμάτων. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι στις προηγούμενες περιόδους ε, το ποσοστό ήταν πάντα πάνω από το 5%, αρκετά πιο πάνω, και η τάση είναι καθοδική και αυτό είναι λόγω του ενισχυμένου ε, μοντέλου διασφάλισης για το 2015-2018. Οι πιστοποιημένοι αιτήσιοι λογαριασμοί και οι έγκαιρες διορθώσεις βοήθησαν πάρα πολύ. Επίσης, με τη στήριξη της Επιτροπής μας ε, ε, συνεργαστήκαμε και με τα κράτη-μέλη για τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και φέτος ε, το ποσοστό είναι υψηλότερο σε σχέση με πέρσι γιατί έχουμε πολύ περισσότερα προγράμματα με επιστοποιημένους λογαριασμούς, 175 σε σχέση με τα 35 πέρσι και αύξηση στις δηλωμένες δαπάνες με περισσότερους εγγενείς κινδύνους και αυτό το ανέφερε και το ελεγκτικό συνέδριο. Φέτος υπάρχει διαφορετική ερμηνεία και αντιλήψη για τους κανόνες, για τα αιτιολογημένα προγράμματα, με πολύ σημαντικό όμως αντίκτυπο για τα σφάλματα τα οποία εκτιμά το δικαστήριο. Οι σχετικές διορθώσεις λοιπόν θα πρέπει να βασίζονται σε κανόνες και σε ε, συγκεκριμένους ε, νομικούς όρους και δεν ισχύει κάτι τέτοιο με αυτά τα σφάλματα. Ε, εάν λάβουμε όμως μέτρα απλοποίησης για να έχουμε ένα σταθερό περιβάλλον, θα συνεχίσουμε να έχουμε τον κίνδυνο αυτών των διαφορών στην ερμηνεία των κανόνων. Για μένα αυτό διακυβεύεται σε αυτή την περίπτωση, η απλοποίηση, αλλά θα πούμε περισσότερα από αυτό αργότερα. Προς το παρόν θα ήθελα να εξηγήσω λίγο την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο στόχος μας σε σχέση με τον κανονισμό είναι ότι τα ποσοστά σφαλμάτων θα μείνουν πει, ε, ε, κάτω από το ποσοστό υλοποίησης ε, ε, για ε, κάθε χρόνο και για κάθε πρόγραμμα. Αυτό γίνεται για να έχουμε εξασφάλιση και να έχουμε τα κατάλληλα προγράμματα που χρειάζεται. Η Γενική Διεύθυνση έκανε έκθεση για κάθε έκθεση και για κάθε ποσοστό σφάλματος, για κάθε ένα από τα 175 προγράμματα το 2018. Επ' αυτής της βάσεως έγιναν και επιτόπου έλεγχοι βάση κινδύνων. Το 2018 έγιναν και πάλι έλεγχοι για ε, επιδειγματοληπτικής βάσεως σε 42 προγράμματα τα οποία θεωρήθηκαν υψηλού κινδύνου και έγιναν αντίστοιχες προσαρμογές. Η έκθεση της Γενικής Διεύθυνση Ρέτζου ανέφερε λοιπόν το ποσοστό σφάλματος και για 175 προγράμματα και είμαστε στο 2 με 3% βάσει μιας διευρυμένης προσέγγισης για κάποια προγράμματα. Παρεμπιπτόντω, ακολουθήσαμε και τη σύσταση του Ελεκτικού Συνεδρίου πέρσι για τον τρόπο υπολογισμού αυτού του ποσοστό σφάλματο. Για να ολοκληρώσω, πιστεύουμε ότι τα στοιχεία μα και η μεθοδολογία μα ε, είναι τα σωστά και μα δίνουν ένα πολύ καλό επίπεδο λεπτομέρειε για να κάνουμε τι απαραίτητε επιπλέον δημοσιονομικέ διορθώσει, ακόμα και αυτέ που χρειάζονται βάσει των ρυθμιστικών εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μα και με την ε, διάθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εξουσία που έχει για τη διαχείριση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Στη συνέχεια, ε, δεν είμαστε μόνο εμείς αυτοί που θέλουμε να εξασφαλίσουμε τα όσα κάνουν ε, είναι και δαπανούμε σωστά τα χρήματα των φορολογουμένων πολιτών. Θα ήθελα να ε, αποτίσω φόρο τιμής στις ελεγκτικές αρχές. Ε, τα εφαρμόζουν πάρα πολύ για πάρα πολλά προγράμματα της περιφερειακής ανάπτυξης σε δύο προγραμματικές περιόδους και είχαμε πάνω από 500 ε, εθνικές εκθέσεις. Είχαμε περίπου 3.300 ε, συναλλαγίες ή τμήματα συναλλαγών που κάλυπταν το 1 τρίτο των δαπανών που δηλώθηκαν σε όλα τα προγράμματα και θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι πρόκειται για μια αναλυτική και εύρωστη βάση, βάση των οποίων μπορούμε να αντλήσουμε συμπεράγματα. Βεβαίω, ε, οι έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνουν και περαιτέρω σφάλματα και ζητούν βελτιώσει σε κάποιε περιπτώσει. Αλλά σε γενικέ γραμμέ θεωρούμε ότι οι αρχέ ελέγχου είναι επαγγελματικέ, ανεξάρτητε και οι περισσότερε από αυτέ εργάζονται βάσει των προδιαγραφών και των προτύπων. Δεν ελέγχουμε μόνο τι ενδιακτικέ αρχέ, και οι διαχειριστικές αρχές και αρχές πιστοποίηση διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για τη δήλωση των δαπανών. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουμε αδυναμίες ή παρατυπίες, απαιτείται και διορθωτική δράση για την βελτίωση των συστημάτων. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι υπάρχει ε, ανάγκη ή περιθώριο βελτίωσης και παρέχεται και τεχνική συνδρομή για συγκεκριμένες ε, ε, ικανότητες. Δίνω και λεπτομέρειες στις απαντήσεις στις γραπτές ερωτήσεις. Όπως βλέπετε λοιπόν έχουμε ένα πλήρες σύστημα και βασιζόμαστε σε στοιχεία από τους ελέγχους και τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς επίσης και πληρωμές για την προστασία ε, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού όπου διαπιστώνουμε ότι είναι ελληματικά τα συστήματα. Δεν ε, θα κλείσει βέβαια το κεφάλαιο της συμμόρφωσης χωρίς να σας επενθυμίσω ότι δεν είναι ε, απάτες οι παρατυπίες. Μόνο το 0,5% ε, είναι υποψία απάτης. Έχουμε μηδενική ανοχή για την απάτη και για όποιον θέλει να εποφοληθεί των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Έχουμε την πρόσφατη έκθεση για την απάτη και τη συνοχή και επιβεβαιώνονται οι βελτιώσει με τα υποχρεωτικά μέτρα τα οποία ισχύουν για κάθε πρόγραμμα. Οποιαδήποτε υποψία απάτη κοινοποιείται στον Όλαφ και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευτεί ο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Ε, δεν διστάζουμε να ζητήσουμε από τις αρχές πιστοποίησης να σταματήσουν τις πληρωμίες ε, ή να επιβάλλουμε διορθωτικές, διορθωτικές πράξεις. Αλλά η να επιβαλλουμε διορθωτικες διορθωτικες αλλα η πολλές παρατυπίες ε, είναι παραβίαση κάποιου άρθρου των κανόνων ή λογοσύνθετων κανόνων. Ε, μπορεί να οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος, ε, σε μείωση, μειωμένες δυνατότητες ε, ή γνώσεις. και πολλά από αυτά θα μπορούσαν να βελτιωθούν με την απλοποίηση. Κάτι το οποίο θα ήθελα να τονίσω εδώ στη συζήτηση είναι ότι η απλοποίηση είναι το βασικό στοιχείο για να μειώσουμε τα σφάλματα και να έχουμε πιο αποτελεσματική διαχείριση και ένα σύστημα ελέγχων και επιθεωρήσεων. Και αυτό είναι η τρίτη μου παρατήρηση. Σύμφωνα με μία μελέτη, οι ε, απλοποίησεις που, εφαρμόστηκαν, που προτάθηκαν συγγνώμη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μειώσουν το διοικητικό κόστος κατά 25% και επειδή μεταξύ των 30 και του 40% των σφαλμάτων που διαπιστώνονται από το ελεγκτικό συνέδριο και από τις ελεκτικές αρχές ε, και από εμά είναι για τις επιλέξιμες δαπάνες, η απλοποίηση είναι πολύ χρήσιμο μέσο για να μειώσουμε τα ποσοστά σφάλματος, καθώς επίσης και η εξοικονόμηση πόρων που θα έλθει και αυτή με την απλοποίηση. Αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι σε όλα τα κράτη-μέλη έχουμε περίπου 2.000 ανθρώπους σε εθνικό επίπεδο που ασχολούνται με τους ελέγχους αυτούς. Ε, εδώ σημαίνει ότι αποκλείουμε και ελεγκτές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και είναι λογική και η απλοποίηση και από διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εκμεταλλευτούν πλήρω τι δυνατότητε που προσφέρει ο κανονισμό, να χρησιμοποιήσουν επιλογέ απλοποιημένου κόστου και θα μειωθεί έτσι το ποσοστό σφάλματο που σχετίζεται με την επιλέξιμη δαπάνη. Επίση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, καταργήσουν του δικού του περιτού κανόνε ε, και πρέπει να ε, δούμε και τις συγκεκριμένε προτάσεις που κάναμε για την επόμενη ε, περίοδο. Υπάρχουν ριζοσπαστικές προτάσεις στον καινούριο κανονισμό και προτείνουν και 80 μέτρα βασικών απλοποιήσεων που θα βοηθήσουν τη μείωση των σφαλμάτων και θα επιταχύνουν την εφαρμογή επιτόπου. Ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία απλοποίησης θα παραμείνει στην τελική συμφωνία διότι η απλοποίηση των κανόνων θα μειώσει και τα ποσοστά σφάλματος, αλλά θα ε, μειώσει και ουσιαστικά και το διοικητικό κόστος και θα εξασφαλίσει και καλύτερη εφαρμογή της πολιτικής. Και έρχομαι στην τέταρτη και τελευταία παρατήρηση, επιδόσεις ε, και αποτελέσματα. Ο βασικός στόχος είναι να υπάρχει αντίκτυπος επιτόπου και να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών. Η συμμόρφωση με τους ε, κείμενους κανόνες είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη και πρέπει να προσέχουμε και τα ποσοστά σαλφαλμάτων, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ε, προσπαθήσουμε να τις μειώσουμε περαιτέρω. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και το γενικότερο πλαίσιο. Η πολιτική για θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και επενδύσεις δεν αρκεί από μόνη της ε, ε, αν πανούμε και μόνον. Πρέπει να κάνουμε στρατηγικές επενδύσεις που θα αλλάζουν ουσιαστικά τις ζωές των ανθρώπων. Για παράδειγμα, μέχρι το τέλος του 2018 η υποστήριξη που δόθηκε σε 300.000 ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υποστηρίζει τη ραχοκαλιά της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη χρηματοδότηση περαιτέρω δυνατοτήτων παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που είναι πολύ περισσότερο από την παραγωγή ενέργειας που είχαμε, για παράδειγμα, στη Λιθουανία. Είναι πολύ εντυπωσιακά τα ποσοστά. Αυτό λοιπόν είναι αυτή η πολιτική. Μόλις ολοκληρώσαμε την ε, εξέταση των επιδόσεων, είδαμε τα προγράμματα και τις προτεραιότητες που λειτουργούν αποτελεσματικά και ποια υστερούν και βάσει αυτών περίπου 3 δις ευρώ από το αποθεματικό ε, διατέθηκαν πλέον σε καλύτερες προτεραιότητες και πέραν αυτών η πολιτική συνοχής δημιουργεί πολλά θετικά αποτελέσματα και στις ε, δημόσιες πολιτικές και στο επιχειρηματικό περιβάλλον και μέσω της εξάντερεσιμότητας. Είναι λοιπόν απτές οι πολιτικές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια. Σας προτρέπω λοιπόν να παρακολουθήσετε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των προγραμμάτων στο απεικαιροποιημένο η πλατφόρμα δεδομένων του ESIF και που έλαβε και βραβείο από τον διαμεσολογητή για την δημόσια διοίκηση το 2017. Τέλος, θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω και το ελεγκτικό συνέδριο με τον κύριο Μέρφυ, καταρχάς και το προσωπικό του για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και για αυτή την ετήσια διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στα μέλη της Επιτροπής, ξεκινώντας από την κυρία Κινίτσι που αντικαθιστά την κυρία Χολμαϊρ, την εισηγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρεμβαίνω εξ ονόματος κυρίας Χολμαϊρ που κολλείεται σήμερα και θα ήθελα και εξ ονοματός της να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο, τον κύριο Μέρφη δηλαδή για την ετήσια έκθεση και τον Επίτροπο τον κύριο Χάν για τις ε, απαντήσεις που έδωσε στις ερωτήσεις μας που είναι οπωσδήποτε χρήσιμες για να ετοιμάσουμε την έκθεση για την απαλλαγή. Για την κυρία Ολμάιρ παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που θα ήθελε να θέσει. Κάποιες από αυτές απευθύνονται προς την Κομισιόν. Η πρώτη από αυτές αφορά τις απαντήσεις σας, οποίες λέτε ότι οι διορθώσεις αυτές παίζουν ένα ρόλο κινήτρου στα κράτη-μέλη για να υποβάλουν εκθέσεις οι οποίες θα είναι κανονικές όμως Υπάρχει μια σειρά αλαθών οι οποίες έχουν ανακαλυφθεί στην δουλειά των κρατών μελών. Μέχρι στιγμή λοιπόν δεν έχει υπάρξει καμία δημοσιονομική διόρθωση. Αναρωτιόμαστε λοιπόν εάν είναι τόσο αυστηρά τα κριτήρια ώστε να μην μπορεί να τα ικανοποιεί κανείς, ποιο ρόλο κινήτρου παίζουν αυτές οι διορθώσεις. Ποιες διορθώσεις έχουν επιβληθεί από την Κομισιόν συνολικά μπορείτε να μας δώσετε μια συνολική εικόνα γραπτός, καθορίζοντας όλες τις δημοσιονομικές διορθώσεις ανά κράτος μέλος. Μετά, για τα προγράμματα τα οποία δεν λειτουργούν αποτελεσματικά κατηγορία 3 και 4. Δυστυχώς η Κομισιόν δεν απάντησε στις ερωτήσεις μας για την ε, πιθανότητα να βρεθεί ένα τέτοιο μοντέλο. Και το περισσότερα από αυτά τα προγράμματα, τα 44 προγράμματα, είναι από την ε, Γαλλία ή την ε, Ουγγαρία. Συνέβαινε αυτό το πράγμα πάντα σε βάθος χρόνου. Γιατί δεν λειτουργούν αυτά τα προγράμματα και γιατί δεν, έχει, δεν έχουν τροποποιηθεί. Θα μπορούσε η την ουγγαρια συνεβαινε αυτο το πραγμα παντα σε βαθος χρονο γιατι δεν λειτουργουν αυτα τα προγραμματα και γιατι δεν εχει δεν εχουν τροποποιηθει θα μπορουσε η κομισιον να μας πει ποιες είναι οι συστάσεις, υπάρχουν παρόμοια προβλήματα σε άλλα προγράμματα. Όσον αφορά τις εθνικές ελεγκτικές αρχές, η απάντηση στην ερώτηση 16 αναφέρει την βελτίωση της κατανόησης των διατάξεων από τις εθνικές ελεγκτικές αρχές και καλύτερη εκπαίδευση του προσωπικού ως τις δράσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν για να βελτιωθεί η αξιοπιστία τους. Βλέπουμε όμως την απάντηση στην ερώτηση 8 πως ε, δεν συμφωνείτε με το ότι η έλλειψη εκπαίδευσης ε, είναι κάτι το οποίο εμποδίζει τις εθνικές ε, αρχές. Μα αν αυτό δεν τις εμποδίζει, ποιες είναι οι βασικές αιτίες των σφαλμάτων στο επίπεδο των εθνικών ελεκτικών αρχών. Και Όπως ήδη ακούστηκε, οι εθνικές ελεγκτικές αρχές ανακάλυψαν 60 σφάλματα. Ε, το λιγότερο από τα δύο τρίτα. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος ε, κατά την άποψή σας. Επίσης, ε, μιλήσατε για την τεχνική αρρωγή. Τα κράτη-μέλη λέτε ότι δεν χρησιμοποιούν επαρκώ τα σχετικά κονδύλια για να βελτιωτήσουν την διοικητική ικανότητά τους. Αν όχι, γιατί. Υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν ιδιαίτερα μικρό ρυθμό απορρόφησης των κονδυλίων της τεχνικής αρχής και τι άποψη έχετε για ένα σύστημα ανταλλαγής δεξιοτήτων στο οποίο οι εθνικοί ειδικοί, ειδικά οι πιο αποτελεσματικοί, θα περάσουν λίγο χρόνο εργαζόμενοι στις αρχές των κρατών που είναι λιγότερο αποτελεσματικές. Θα μπορούσε ένα τέτοιο σύστημα να είναι λειτουργικό και να εισαχθεί. Και θα μπορούσε να κάνει κομισιόν ε, σχετικά. Επίσης, τι θα κάνει η Κομισιόν για να υπάρξει μια διαρκής βελτίωση της απόδοσης των εθνικών ελεγκτικών αρχών. Και κατόπιν κάποιες ε, ερωτήσεις για το ποσοστό απορρόφησης. Ε, δεδομένου του ότι σε πολλές χώρες της ε, συνοχής το ποσοστό αυτό είναι χαμηλό. Οφείλεται αυτό στην έλλειψη διοικητικής κανότας και συγκεκριμένα στην ε, δυνατότητά τους να υποστηρίξουν τους ε, υποψηφίους και κάτι ακόμα. Υπάρχουν ε, κάποια κράτη-μέλη στα οποία το μεγαλύτερο μέρος των δικαιούχων λαμβάνει κυρίως κονδύλια της συνοχής ή εκεί πέρα τα κονδύλια συνοχής φτάνουν σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων. Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μια ουδέτερη αξιολόγηση των υποψηφιωτήτων σε σχέση με τους ε, δικαιούχου. Και τέλος κάποιε ερωτήσει για το ελεγκτικό συνέδριο. Θα ήθελα λοιπόν ε, να σας ρωτήσω για την τεχνική αρρωχή, πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η τεχνική αρρωχή και η ανταλλαγή των ε, βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών ελεγκτικών αρχών. Έχει υπάρξει κάποια βελτίωση τα τελευταία χρόνια και με βάση τις απλοποιήσεις οι οποίες αναφέρθηκαν θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι τέτοιο στο επίπεδο των κανόνων. Τέλος, όσον αφορά την περίοδο 2014-2020, είχαμε ένα επίπεδο σφαλμάτων υψηλότερο από την περίοδο την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Επίσης η Κομισιόν αναφέρθηκε στο ελεγκτικό συνέδριο. Το ελεγκτικό συνέδριο είπε πως ε, τα κράτη-μέλη έχουν, υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που έχουν ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανομαλιών. Αυτά και σας ευχαριστώ και εγώ και η κυρία Χολμαϊρ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, η σκιώδης εισηγητές, η κυρία Πίνκοβα από τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ το Ελληνικό Συνέδριο για την λεπτομερή έκθεση. Ε, ευχαριστώ τον κύριο Μέρφυ για την παρουσίαση. Ευχαριστώ επίσης Επίτροπε Χάν για την εισηγησή σας και τα σημεία που τονίσατε σε αυτήν. Έχω τρεις ερωτήσεις που θα ήθελα να ε, σας απευθύνω. Η πρώτη αφορά τον κανονισμό για την πολιτική συνοχή στον οποίο αναφερθήκατε ότι επέτυχε πολλά. Ξέρω πως σύντομα εξηγήσατε τους τομείς ε, τους οποίους ορίζεται επιτυχής, αλλά μπορείτε να μας μιλήσετε για συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία επιτόπου εντοπίζεται ως επιτυχή. Η δεύτερη ερώτηση έχει δύο τμήματα και ε, σχετίζεται με τον προσανατολισμό του προγράμματος και την εισαγωγή του αποθεματικού απόδοσης ε, το 2019. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού του αποθεματικού ε, απόδοσης και επίσης δεν συνεχίζεται αυτό στην προγράμματα της νέας γενιάς. Αυτό σημαίνει πως ε, η απόδοση θα θυσιαστεί προς όφελος της απλοποίησης του κανονισμού ή τι προβλέπετε. Αυτό ήταν το δεύτερο κομμάτι της δεύτερης ερώτησης. Και το τελευταίο, η τελευταία ερώτηση αφορά κάτι που είχε, ήδη είχε θυγεί από την κυρία Χολμάγερ, αλλά θέλω να μια περαιτέρω διευκρινήση και είναι το πώς εξασφαλίζεται την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων στις νομοδοτήσεις που εκδίδουν οι ελεγκτικές αρχές. Εφόσον υπάρχουν πάνω από 126 διαφορετικές αρχές, μπορείτε να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες για την διαδικασία αξιολόγηση της εργασίας των διαφόρων αυτών αρχών, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στον κύριο Σαστέλα από το Ρηνιού. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θέλω και εγώ βεβαίως να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση της έκθεσης δραστηριοτήτων ε, ε, για την περιφερική πολιτική που συμπληρώνει την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου, το οποίο και ευχαριστώ επίσης για την εργασία του. Για την γάμα δέλτα οι δείκτες τη απόδοσης είναι σημαντικοί, διαγνωρίζοντας ότι η συνοχή αντιπροσωπεύει πάνω από 54 δις, δηλαδή δηλαδή 35% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Και όσον αφορά τα ποσοστά σφάλματος και το συζητήσαμε, το ποσοστό σφάλματος από την Κομισιόν για την συνοχή, η ετοιμιγορία στα μάτια του δικαστηρίου είναι αδιαφεσβήτητη γιατί θεωρεί πως δεν μπορεί να το εμπιστευτεί γιατί μάλιστα αναφέρει ε, διαρκείς αδυναμίες όσον αφορά την κανονικότητα των δαπανών που αναφέρονται από τις αρχές διαχείρισης. Έλλειψη αξιοπιστίας των στοιχείων που δίνουν τα κρατημέλη και είναι ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα και μάλιστα είναι ε, επίμονο το πρόβλημα αυτό και επαναλαμβάνεται. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει αφιβολίες. 13 αρχές ελέγχου έχουν αναφέρει ε, μόνιμο σφάλμα κάτω του 2% ενώ το ελληνικό συνέδριο εκτιμά πως είναι γύρω στο 5%. Πώς ε, μπορεί οι εθνικοί οργανισμοί ελέγχου να μην ανοιχνεύουν σφάλματα ενώ το ελεγκτικό συνέδριο μπορεί να τα εντοπίσει. Πώς θα διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Έχουν γίνει επαφές με τα κατημέλη που ε, ε ορίζουν επιπλέον κανόνες και έτσι καταστούν ακόμη πιο περίπλοκη τη διαδικασία και άρα τον κίνδυνο σφάλματος. Το ελεγκτικό συνέδριο αναφέρει στοιχεία ε, και διευκρινίζει ότι μπορούμε πάντοτε να μην εμπιστευόμαστε ε, το ποσοστό σφάλματος και πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτές τις κρίσιμες και βασικές επικρίσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, το οποίο ε, προτείνει κάποιες συστάσεις. Αυτές θα εφαρμοστούν. Ε, ποια συνέχεια θα δοθεί. Επίσης, το συνέδριο ε, επιμένει ε, όσον αφορά τον αντίκτυπο του σφάλματος, ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να ενημερωθούν οι ετούντες για τους ισχυοντές κανόνες. Επιπλέον, ποια είναι τα μέτρα που προβλέπονται ώστε να διευκολυνθεί και να ενταθεί η απορρόφηση του προϋπολογισμού ώστε να υπάρξει πραγματική οικονομική οικονομική ανάπτυξη πιο σημαντική από αυτή που παρατηρούμε. Ε, επίσης, το Ελληνικό Συνέδριο επικρίνει τους δείκτες απόδοσης που χρησιμοποιούνται ε, επί τη βάση του ότι αυτοί οι δείκτες αποτελεσμάτων δεν είναι πάντοτε κομμάτι της ίδιας της ε, σύλληψης των προγραμμάτων. Αυτά λοιπόν τα προγράμματα θα αναθεωρηθούν. Τι συμβαίνει με τα κράτη-μέλη όπου πολλά από αυτά δεν έχουν δείκτες ή έχουν εν πάση περιπτώσει δείκτες που δεν αποδίδουν. Ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πίξα από τους Πρασίνους. Θα μιλήσω τσεχικά. Σας eh, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας μιλήσω. Θα μιλήσω για την ε, κοινή διαχείριση. Θεωρείτε ότι τα κράτη-μέλη θα ελέγχουν εαυτούς. Τι ε, διασφάλιση υπάρχει όταν ε, έχουμε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη ή όταν έχουμε συγκρόμνα συμφέροντα όπως την Τσεχία και όταν έρχονται κάποια πράγματα στο φως όπως λένε οι Τσέχοι και οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι τι θα κάνετε για να προστατεύσετε τα ευρωπαϊκά κονδύλια από πολιτικούς όπως ο Αντρέι Μπάμπης και ο Βίκτορ Όρμπαν Σας ευχαριστώ θα το, λόγο. θα πάρει τώρα ο κύριος Χάνα για να απαντήσει σε όλες αυτές τις παρεμβάσεις. Thank you very much. I think... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω σε γενικές γραμμές υπάρχουν κάποια ζητήματα. Ένα αφορά την μεθοδολογία. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ των όσων κάνει το ελεγκτικό συνέδριο και εμείς. Αλλά αυτό το οποίο κάνουμε εμείς και οι εθνικές αρχές είναι να κοιτάμε σχεδόν την κάθε συναλλαγή. Και αν το συγκρίνετε, είναι σαν να το συγκρίνετε με ένα γκάλοπ. Δηλαδή αν ρωτήσουμε 2-3 άτομα θα έχουμε ένα πολύ μικρό φάσμα αποτελεσμάτων. Εάν έχουμε ένα δείγμα ατόμων, το φάσμα είναι τελείως διαφορετικό. Και αυτή είναι μια εξήγηση ε, για τις διαφορές αυτές. Αλλά υπάρχει κάποια επικάλυψη. Ε, θα έλεγα ότι το δικό μας ποστό σφάλματος είναι στο κάτω όριο του σφάλματος ε, του δικαστηρίου, οπότε δεν βλέπω κάποια μεγάλη διαφορά. Θα έλεγα ότι είναι το αποτέλεσμα διαφορετικής μεθοδολογίας. Δεύτερον, αν έχουμε ενδείξεις ότι η δουλειά των ελεγκτικών αρχών ε, δεν είναι τέλεια, ε, θα το δούμε. Και δεν βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη τάση όπου κάποιες χώρες έχουν μόνιμες αδυναμίες και βεβαίως η κατάσταση είναι διαφορετική από όταν ήμουν Επιτροπός Συνοχής πλήρους απασχόλησης, αν μου επιτρέπετε, γιατί τότε δύο χώρες κάθε χρόνο είχαν πρόβλημα στον έλεγχο, κάτι το οποίο μεταξύ διορθώθηκε με εντατική εκπαίδευση και όλα τα σχετικά. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει μια βελτίωση και θυμάμαι πολύ καλά ότι όταν έφυγα ε, πριν από πέντε χρόνια δεν θεωρούσα ότι είναι δυνατόν να έχουμε καλύτερο ποσοστό σφάλματος από το 5% αλλά ε, από ό,τι φαίνεται είναι. Νομίζω ότι όλοι πετύχαν πολλά αλλά είναι και θέμα του να βρεθεί η σωστή ισορροπία. Ε, Τώρα αναφέρθηκα στον μεγάλο αριθμό ανθρώπων που ασχολούνται με την ετήσια διαδικασία ελέγχου και νομίζω ότι Έχουμε και το όριο σημαντικότητας. Κάτι το οποίο θεωρώ ένα τεράστιο επίτευγμα. Νομίζω λοιπόν ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες και πάλι αν έχουμε περισσότερη απλοποίηση κίνδυνος, το επίπεδο των δυνητικών κινδύνων πέφτει, γιατί όπως σας είπα ένα 50% των σφαλμάτων σχετίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με την διαφορετική ερμηνεία της επιλεξιμότητας ε, των δαπανών και αυτό οφείλεται και στην ε, περιπλοκότητα. Σε πολύ ε, μικρά έργα. Γι' αυτό προτείναμε για τον επόμενο κανονισμό την εισαγωγή ποσών ε, καταποκοπήν και απλοποιημένου κόστους για έργα μέχρι 200.000 ευρώ. Έτσι ώστε οι δικαιούχοι που δεν είναι λογιστές να μπορούν να εφαρμόσουν τους κανόνες και να αποφεύγουν τα λάθη. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει συμμεθεί σημαντική πρόοδος και νομίζω ότι μπορεί να γίνουν περισσότερα. Και αν μου επιτρέπετε να μιλήσω με τη μελλοντική μου ιδιότητα ως Επίτροπος ε, και για την εσωτερική ψηφιοποίηση, τη ζήτησα από το προσωπικό εάν μπορεί να δει την δυνατότητα διαλειτουργικότητας μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και διαχειριστικών και ελεγκτικών αρχών στα κράτη-μέλη. Και να δούμε ακριβώς την εφαρμογή των έργων εγκαίρως και να αποκλείσουμε τα περαιτέρω σφάλματα για να έχουμε ένα σύγχρονο ελεγκτικό σύστημα και με στήριξη της πληροφορικής. Μια εξαιρετική ιδέα της κυρίας Χόλμα και άλλων είναι αυτή η ανταλλαγή δεξιοτήτων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Και υπάρχει νομίζω δυναμικό που δεν έχουμε εκμεταλλευτεί μεταξύ των ελεγκτικών αρχών και της Κομισιόν και των διαχειριστικών αρχών. Και αν μου επιτρέπετε θα έλεγα και στο ηλεκτρικό συνέδριο. Και ελπίζω να μπορεί να εφαρμοστεί το... ο λόγος για τον οποίο έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην απορρόφηση. Οπωσδήποτε σχετίζεται με πολλά θέματα. Ένα από αυτά είναι Οπωσδήποτε και γι' αυτό θέλουμε ακριβώς να έχουμε συμφωνία στο επόμενο ΠΔΠ. Γιατί βλέπουμε ότι η απόφαση αυτή έχει δημιουργήσει καθυστερήσεις. Δεύτερον, η εισαγωγή του ΝΙΣΙΝΤΡΙΑ 3 δεν έχει συνεισφέρει σε πιο αποτελεσματική εφαρμογή, έχει οδηγήσει σε επανάπαυση. Και τέλος, για πρώτη φορά έχει εισαχθεί εδώ η ανάγκη για κάθε κράτος μέλος να προκύψουν κάποιες στρατηγικές, παραδείγματος χάρη μεταφορές Θυμάμαι λοιπόν όταν είχα ξεκινήσει το 2010 αντιμετώπιζα άχρηστα αεροδρόμια, λιμάνια ανά την Ευρώπη. Ε, πλέον αυτό δεν είναι ζήτημα γιατί εντωμεταξύ έχουμε επιβάλει μια ολιστική στρατηγική σε ολόκληρη την χώρα. σε όλα τα μέσα μεταφοράς και πρέπει να πω ότι σε κάποιες χώρες χρειάστηκε χρόνος για να απτυχθεί μια τέτοια στρατηγική. Αλλά οπωσδήποτε έχει βελτιωθεί η ποιότητα των ε, έργων και νομίζω ότι μπορούμε στην επόμενη περίοδο να βασιστούμε σε όλα αυτά. και έχουμε ξεκινήσει κάτι το οποίο οπωσδήποτε θα αποδώσει ε, στην επόμενη περίοδο. Υπήρξαν κάποιες συζητήσεις για την ε, εξέταση αυτή της απόδοσης. Και ε, μπορώ να σας πω ότι η έκθεση έδειξε ότι οι συνολικές δραστηριότητες είναι γύρω στο 75% του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και το αποθεματικό των Ταμείων Συνοχής ε, είχαμε ένα 90% και 75% ε, για το ΕΤΠΑ και έχουμε 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία πηγαίνουν σε στόχους που αποδίδουν αλλά 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το αποδηματικό συνδέεται με προτεραιότητες που δεν πέτυχαν τα ορόσημα απόδοσης. Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να προταθεί μια ανακατανομή και αναλύουμε προσεκτικά όλα αυτά τα πράγματα. Η επόμενη εξέταση θα γίνει το 2024 για τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό είναι λοιπόν το πρόγραμμα. Κάποιος άλλος με ρώτησε για κάποια πολύ καλά παραδείγματα αν παρακολουθείτε τα βραβεία Regio Stars, θα δείτε το πώς πηγαίνουν τα διάφορα έργα, καμιά φορά μικρά, άλλες φορές μεγάλα. Και νομίζω ότι εδώ πέρα βλέπουμε την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Νομίζω έχουμε πετύχει πάρα πολλά πράγματα με ψηφιακό μετασχηματισμό σε διάφορες χώρες για διάφορους στόχους, διασυνοριακά έργα σε Γαλλία και σε Benelux όταν μιλάμε για τη βιώσιμη κατανάλωση, τα έξυπνα δίκτυα και πολλά άλλα θετικά παραδείγματα. Είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος μας δείχνει ότι η πολιτική συνοχή είναι μια πολύ σύγχρονη πολιτική ε, και ακριβώς αυτή είναι η ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πετύχει συγκεκριμένους στόχους και θα το δείτε αυτό στην επόμενη περίοδο όταν ε, ένα 30% των κονδυλίων συνοχής και περιφερειακών των ταμείων θα πάει σε κλιματικές δράσεις και τα σχετικά για να επιτύχουμε τις πολιτικές μας ε, προτεραιότητες. Το ίδιο ισχύει και για τον ψηφιακό κλάδο. Τώρα, αν ξέχασα κάτι, θα απαντήσουμε γραπτός. Για τον συνάδελφο από την Τσεχία, αν υπάρχουν ενδείξεις κατάχρησης, ε, σταματάμε τις πληρωμές και το έχουμε ήδη κάνει. Στις περιπτώσεις που αναφέρατε λοιπόν έχουμε σταματήσει τις πληρωμές. Δεν υπάρχει κάποια ε, ζημία λοιπόν που υφίσταται ο Ευρωπαίος φορολογούμενος, αλλά υπάρχουν και άλλοι έλεγχοι. Και αυτό αφορά και εθνικούς κανόνες. Και βεβαίω ε, θα έρθει αρχές Δεκεμβρίου, θα έρθουν οι σχετικοί κανόνες, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και στοιχεία για τις επιτυχίες αυτές, ε, τουλάχιστον και με των θερών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Και ε, δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει και ο κύριος Μέρφη στις ερωτήσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ναι. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον ε, τις ερωτήσεις ε, και τα σχόλια των ομιλητών και τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που έθιξαν. Όσον αφορά τις συγκεκριμένε ερωτήσεις προς το ελληνικό συνέδριο, νομίζω κυρίως τις έκανε η κυρία Κινίτσεκ εκ μέρους της κυρίας Χολμαϊερ. Όσον αφορά την τεχνική συνδρομή, νομίζω συμφωνώ με τα όσα είπε ο ε, Επίτροπο για την ανταλλαγή δεξιοτήτων. Είναι καλή ειδικία και πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί πολύ για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Υπάρχουν πάρα πολλέ ομάδες εργασία, τι οποίες συμμετέχουμε και εμεί ως παρατηρητές ε, σε κάποιες και ε, έχουν γίνει προσπάθειες για την βελτίωση της κατάστασης. Νομίζω ότι τα συνόψισε εξαιρετικά ο Επίτροπος Χάν. Είναι πολύ σύνθετος ο τομέας και είναι πολύ δύσκολο να έχουμε την ίδια προσέγγιση για όλα τα κράτη-μέλη. Αναφέρθηκα στο γεγονός ότι τον εξέπληξε, ε, ότι δεν θα είχε φανταστεί ότι θα είχαμε ποσοστό σφάλματος του 5%. Είναι καλό το ότι φτάσαμε σε αυτό, αλλά νομίζω ότι η φύση των συναλλαγών είναι τέτοια και τόσο σύνθετη που ε, σημαίνει ότι πρέπει απλώ να προσπαθούμε να παρέχουμε τεχνική συνδρομή και η πρόοδο θα έρθει, αλλά είναι αργή η διαδικασία. Όσον αφορά την απλοποίηση των κανόνων, εμεί είμαστε αναφανδόν υπέρ τη απλοποίηση. Το έχουμε πει επανειλημμένω ότι υπάρχουν ε, δυνατότητε ε, απλοποιημένου κόστου και όπου χρησιμοποιούνται έχουμε μικρότερο ποσοστό σφάλματο, αλλά βλέπουμε ότι είναι πολύ περιορισμένη η χρήση και αυτό είναι και λίγο απογοήτευση. Επίσης σημειώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, υποβάλει 80 προτάσεις απλοποίησης για την επόμενη περίοδο και τον επόμενο κανονισμό. Έχουμε κάνει και εμείς κάποιες προτάσεις. Ε, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία. Δεν θέλουμε απλώς απλοποίηση για να υπάρχει απλοποίηση. Ορισμένες φορές πρέπει να υπάρχει ε, και έλεγχος σε κάποιες πτυχές και δεν θα πρέπει να χαθεί αυτό. Ρωτήσατε κατά πόσον υπάρχει διαφορά μεταξύ των 26 τομέων στους οποίους διαπιστώσαμε σφάλματα. Υπάρχει. Για το 2007-2013 είχαμε διαπιστώσει 10 σφάλματα σε 5 κράτη-μέλη και για το 2014 2020 ήταν 26 σε 8 κράτη-μέλη. Και όπως λέμε και στην παράγραφο 6 σημείο 14, η συχνότητα από το 2014 στο 2020 ήταν ε, μεγαλύτερη. Γιατί κάποια κράτη-μέλη έχουν σφάλματα και κάποια άλλα όχι. Όπως βλέπετε επισκεφθήκαμε 15 κράτη-μέλη σε αυτό το έτος ελέγχου. Διαπιστώσαμε κάποια σφάλματα σε σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη. 11 κράτη-μέλη καλύπτονται από αυτά τα 26 σφάλματα δεν μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα για ένα κράτο μέλη. Αυτό είναι ένα τυχαίο δείγμα που παίρνουμε για να έχουμε μια εικόνα για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό συνολικά. Δεν παίρνουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα βάσει το οποίο μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για ένα κράτο μέλο. Εξαρτάται από το δείγμα και από τα κράτη-μέλη που περιλαμβάνονται στο δείγμα. Για το 2019 έχουμε προσθέσει άλλα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουμε ακόμα επισκεφθεί η ιδέα είναι να επισκεφθούμε και τα 27 ή 28 κράτη-μέλη μέσα σε ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ένα δεύτερο γύρο παρεμβάσεων τώρα. Η κυρία Τσέ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε στην αξιολόγηση του προπολογισμού θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο να δούμε τα κονδύλια που δαπανάηθηκαν, αλλά και την αποτελεσματικότητα της δαπάνης. Το Μάρτιο του 2018, ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ρέγγιου παρουσίασε αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής για τις τέσσερις χώρες Βίσεγκραντ και τόνισε ότι η Ουγγαρία συστηματικά λαμβάνει τα περισσότερα κονδύλια σε σχέση με το ΑΕΠ της, σε σχέση με την Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία ή τη Σλοβακία. Παρά το γεγονός ότι λαμβάνει τα περισσότερα κονδύλια, θεώρησε ότι η Ουγγαρία, και το τονίζω, έχει πολύ χειρότερε επιδόσει σε σχέση με όλε τις υπόλοιπε χώρε και αυτό για όλου του δείκτε. Ε, για την ανάπτυξη του ΑΕΠ, το ποσοστό τη ε, φτώχεια ε, και άλλου δείκτε. Ποια είναι η ιδέα σα λοιπόν για τη θετική εξόλυξη. Η χώρα που λαμβάνει την περισσότερη χρηματοδότηση και επωφελείται λιγότερο. Θεωρείτε ότι υπάρχει ακόμα αυτό το πρόβλημα και αν ναι, τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον για να βελτιωθούν τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέξα θέλει και πάλι το λόγο. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να θέσω μια επιπλέον ερώτηση. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι σε περίπτωση που υπάρχει συστηματική παρατυπία, σταματάτε τις πληρωμές. Βάσει των πληροφοριών που έχω εγώ, η Agrofed, που είναι η διοκτησία του Τσέχου Πρωθυπουργού, του Ανδρέη Μπάμπιτς, εξακολουθεί να λαμβάνει χρηματοδότηση, παρά το γεγονός ότι αυτό καταβάλλεται από τις τσεχικές αρχές. Αυτό ε, στρεβλώνει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και εγώ θα περίμενα παρέμβαση της Κομισιόν. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουν ληφθεί κάποια μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, μπορείτε να απαντήσετε παρακαλώ και στις δύο παρεμβάσεις. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση για την Ουγγαρία και το γεγονός ε, ότι σε όλα τα σχετικά οικονομικά στοιχεία η Ουγγαρία είναι η πιο αδύναμη σε σχέση με τους άλλους τρεις, ε, ειλικρινά πρέπει να σας πω ότι δεν γνωρίζω το θέμα αυτό, δεν μπορώ να απαντήσω. Αν ε, αναλογιστεί κανείς τα στοιχεία απασχόλησης είναι κάτι το οποίο πρέπει να δείτε από χρονιά σε χρονιά. Δεν ε, ε, μπορώ να σας πω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Uh, Επίσης να πω ότι ε, δεν διακόπτουμε τις πληρωμές μόνο όταν υπάρχει συστηματική κατάχρηση, αλλά και όταν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη περίπτωση, για παράδειγμα, τότε αναστέλλονται αμέσω οι πληρωμές. Εσείς αναφέρεστε σε κάτι άλλο. Αναφέρεστε στην επιδότηση της γεωργικής πολιτικής για τον πυλώνα 1. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει σχέση ε, με μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Αφορά την ε, χρήση ε, της γης, ε, τα σχετικά εκτάρια και οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό και την ιδιοκτησία της γης. Από ό,τι γνωρίζω όμως υπάρχει ένας έλεγχος σε εξέλιξη, αλλά αυτή είναι διαφορά μεταξύ συνοχής και πρώτου πυλώνα στη Γεωργία. Ευχαριστώ πολύ. Για να ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να δώσω και πάλι το λόγο στην κυρία Κινίτσι, αν θέλει να προσθέσει κάτι ακόμα, κάποια παρατήρηση, για να κλείσει αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα απλώς ε, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Επίτροπο Χάν και τον κύριο Μέρφη για τις απαντήσεις που έδωσε στις ε, πάρα πολλές και πρέπει να πω πολύ σύνθετες σε κάποιες περιπτώσεις ερωτήσεις που έθεσα και εγώ εξ ονόματος της κυρίας Χολμάιερ αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Και σας ευχαριστώ και πάλι για τη δέσμευσή σας για να δώσετε περαιτέρω πληροφορίες για τα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν όλους σας το ελεγκτικό συνέδριο τον κύριο Μέρφυ, τον Επίτροπο για τη συζήτηση αυτή, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Και κύριε Επίτροπε, όπως ε, είπατε και στην προηγούμενη παρέμβασή σας, ε, θα είναι η τελευταία συμμετοχή σας τουλάχιστον ως αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας και τη βοήθειά σας και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Είμαι βέβαιη ότι θα σας ξαναδούμε εδώ, αλλά με διαφορετική ιδιότητα θα, ήσασταν, θα είστε Επίτροπος για Προπολογισμό και Διοίκηση. Σας ευχαριστώ και εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρία της Επιτροπής. Mañana. Αύριο μην ξεχάσετε να φέρετε τις κάρτες ψηφοφορίας, γιατί στις 9 η ώρα θα ψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ.